Καλησπέρα σα, κύριε και κύριοι. Καλησπέρα και στα γαλλικά και στα αγγλικά. to... Θα ήθελα παρακαλώ την προσοχή σας για λίγο με τις ανακοινώσεις του Προέδρου για να ξεκινήσουμε ολοταχώς. Αλλά συγκρίνουμε πρώτα τη σε διάταξη αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Please, if you may have your seats so that we can be sure that everyone is ready. Παρακαλώ καθίστε. Γιατί σκοπεύω να αρχίσω καλωσορίζοντα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μία ομάδα βουλευτών από την Αρμενική Βουλή που επισκέπτεται σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλώς ήρθατε Καλωσορίζουμε το κλιμάκιο της Αρμενικής Βουλής. Καλώς ήρθατε μέλη της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που βρισκόσαστε μαζί μας σήμερα. Συνεχίζουμε με τον ορισμό των, των εισηγητών. Η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου θα αναλάβει την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Ο κύριος Λουί Μισελ των Φιλελευθέρων θα αναλάβει την έκθεση για την τροποποίηση του κανονισμού που προβλέπει τον κώδικα, Ευρωπαϊκό Κώδικα Επιχειρήσεων. Και η κυρία Ρενάτε Βέβερ ε, και θα αναλάβει την έκθεση για την ε, αποκατάσταση των ε, ελέγχων στα σύνορα σε εξαιρετικέ περιπτώσεις και η κυρία Ρενάτε Βέμπερ θα συντάξει την έκθεση και για την ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη και τις προδιαγραφέ για, τα... για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία στα μέσα μαζική ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. συμφωνούμε με το διορισμό των εισηγητών. Και περνάμε στο σημείο 3 και 4 που θα εξεταστούν σε κοινή συζήτηση. Καταρχήν να καλωσορίσω και πάλι στην Επιτροπή μας την κυρία Φρανσουάς Λεμπάι τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την κοινή συζήτηση αυτών των δύο σημείων, των σημείων 3 και 4 όπως σας είπα, να σας υπενθυμίσω και την ψηφοφορία που θα γίνει αργότερα. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι αργότερα θα ψηφίσουμε, γι' αυτό φροντίστε, αν δεν έχετε φέρει μαζί τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας, να στείλετε κάποιον να σας τη φέρει να σας τις φέρουν, γιατί θα τις χρειαστείτε αργότερα. Κοινή συζήτηση το σημείο 3 και 4. Δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και δικαίωμα επικοινωνία μετά τη σύλληψη. Και σημείο 4. Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Θα ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση από την κυρία Λεμπάη, τη Γενική Διευθυντήρια Δικαιοσύνη, και μετά θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Θα θυμάστε ότι οι δύο πρωτοβουλίε αφορούν τον οδικό χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2009 το Συμβούλιο μετά την έγκριση τη οδηγία για το δικαίωμα σε διερμηνία και μετάφραση σε ποινικέ δίκε καθώς και την πρόταση οδηγίας για το δικαίωμα ενημέρωσης σε ποινικέ δίκες που βρίσκεται υπό εξέταση αυτή τη στιγμή. Το σημείο 4 εντάσσεται στο πακέτο προστασίας των θυμάτων. Είναι συναφής με την προηγούμενη πρωτοβουλία, πολύ σημαντική και περιλαμβάνει και μία ανακοίνωση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για μια οδηγία που προβλέπει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων και ένα κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασία σε αστικέ υποθέσει, που συμπληρώνει το λεγόμενο πακέτο για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία σε ποινικά θέματα την οποία εγκρίναμε και μάλιστα με ομοφωνία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και πολύ πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα. Θα ακούσουμε, επαναλαμβάνω, την παρουσίαση των δύο σχεδίων εκθέσεων. Αφού ακούσουμε φυσικά την παρουσίαση της κυρίας Λεμπάγη. Μετά θα γίνει συζήτηση. As, ε, ε, for the first report on access to lawyer and criminal... Παραλαμβάνε πρώτη έκθεση αφορά το δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Η συγκήτρια είναι η κυρία Αντωνέσκου και για το πακέτο που αφορά τα θύματα. Η συγκήτριά μα είναι η κυρία Τερέσα Χιμένε Μπεσερίλ. Μπουσουτήλ διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. According to my agenda, we should first be discussing... Το σημείο 3 θα έλεγα να εξετάσουμε πρώτα ε, και ξεχωριστά σε κοινή συζήτηση τα σημεία 4 και 5. Κατάλαβα καλά γιατί κατά τη γνώμη μου τα δύο συναφή θέματα είναι το 4 και το 5, όχι το 3 και το 4. Πιστεύω ότι το 3 θα πρέπει να το εξετάσουμε ξεχωριστά το θέμα δικαίωμα, δικαιώματος πρόσβαση σε δικηγόρο. Ναι, όντω, όντω δίκιο έχετε, λέει ο πρόεδρο. Όντω. Point, point number four. Όντως, τα σημεία 4 και 5 είναι αλληλένδετα. Άλλωστε, αρμόδια για την παρουσίαση και στα δύο θέματα είναι η κυρία Λεμπάιχ. Αλλά το πρώτο θέμα, το 3, που αφορά δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, είναι κάτι ξεχωριστό. Α γίνει πρώτα λοιπόν η παρουσίαση και η συζήτηση για το 3 και κατόπιν σε κοινή συζήτηση θα εξετάσουμε τα 4 και 5. Κυρία Λεμπάγη, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πραγματευτώ το πρώτο θέμα της μέρης διάταξης. Είναι μόνο το πρώτο κομμάτι της ατζέντα, αλλά από ό,τι κατάλαβα θα περάσουμε το απόγευμα παρουσιάζοντα πρωτοβουλίε τη Γενική Διεθνή Δικαιοσύνη, που είναι και δείγμα τη δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αυτά. Το πρώτο θέμα συνδέεται με τα θέματα πρόσβασης ε, σε δικηγόρο. Και όπως είπατε, είναι το διαδικαστικό δίκαιο το οποίο έχουμε υιοθετήσει, που έχει ήδη αποφασιστεί, που είναι ευρία τη ερμηνεία. Το συζητάμε και ευελπιστούμε να ολοκληρώσουμε σύντομα το θέμα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην πληροφόρηση και περνάμε σε αυτό που κατά τμήριο είναι η πιο ενδιαφέρον κομμάτι, που είναι η πρόσβαση σε δικηγορική αρρωγή. Στο θέμα αυτό λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καθορίσουμε τα ελάχιστες προδιαγραφές για ελάχιστες εγγυήσει εξασφάλισης ε, συνηγόρου για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να επιτύχουμε είναι η μετάφραση σε οδηγία ουσιαστικά της ε, νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου που ορίζει ότι θα πρέπει να είναι παρόν συνήγορος από την πρώτη ανάκριση κάποιου υπόπτου από την αστυνομία. Το δικαστήριο του Στρασβούργου υπήρξε σαφές επί του θέματος και υπήρξε εξίσου σαφές ότι το δικαίωμα υπεράσπισης α, αποτελεί πρόκριμα όταν γίνονται δηλώσεις χωρίς παρουσία συνηγόρου ε, και υπάρχει παρεπόμενη καταδίκη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο στοιχείο το οποίο προτείνουμε στην οδηγία αυτή, την απαραίτητη δηλαδή παρουσία συνηγόρου από την πρώτη στιγμή και την πρώτη ε, περίπτωση ανάκρισης υπόπτου. Φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική η έννοια του υπόπτου. Πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί τι κάνει ο συνήγος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε δηλαδή είναι ένας ε, δικηγόρος, ένας συνήγορος που θα είναι δραστήριος, που θα έχει τη δυνατότητα να, να, να μιλήσει κατηδίαν με τον πελάτη του, που μπορεί να είναι παρόν και στην ανάκριση της αστυνομίας ή από άλλες αρχές, που θα έχει το δικαίωμα να θέσει ερωτήματα και να ζητήσει διευκρινήσεις ε, όποτε κρυθεί απαραίτητο. Αυτό που θα θέλαμε λοιπόν να δούμε είναι ένας δικηγόρος που θα είναι δραστήριος, ε, όχι παθητικός, όταν θα παρίσταται για να ε, παράσχει βοήθεια στον πελάτη του. Βέβαια, Εξίσου σημαντικό θα είναι να του δίνετε δυνατότητα να συνδιαλέγεται με τον πελάτη του οποτεδήποτε παρουσιάζονται νέα πιστήρια νέας μαρτυρίας. Για παράδειγμα, ε, σε περίπτωση κατοίκων έρευνε. Ορισμένες φορές για λόγους κατεπήγοντες, όταν για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται κάποιος ε, ε, είδους αναλυτής ή όταν ε, οι μαρτυρίες στοιχειοθετούν ε, κατηγορία. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ των συγκρουόμενων συμφερόντων, μεταξύ του δικαιώματος υπεράσπισης δηλαδή και της ανάγκης διεξαγωγής ανάκρισης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Γι' αυτό και η πρόταση να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να παρεκκλίνουν για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα από το δικαίωμα, από τη θέσπιση του δικαιώματος ε, ε, δικηγορικής ε, αρρωγής όταν υπάρχει κίνδυνος, ιδιαίτερα δημόσια ε, τάξη και ασφάλεια. Όταν όμως ισχύσει η παρέκκληση αυτή, όταν ισχύει η παρέκκληση αυτή, ε, η ισχύση συγγνώμη αυτής της παρέκκλησης θα πρέπει να είναι σε πολύ περιορισμένο διάστημα, για περιορισμένο διάστημα και σε περιορισμένες περιπτώσεις. Μια άλλη σημαντική ε, παράμετρος της προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο παράγων της εμπιστευτικότητας μεταξύ πελάτη και δικηγόρου. Αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση δίκαιας ε, ακροαματικής διαδικασίας στις δημοκρατικές κοινωνίες και βέβαια προφανώς αποκλείει το να είναι ανοιχτό σε μια γενικευμένη παράκαμψη. Και η σύνδεση μεταξύ αυτής της πρότασης και της ε, συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ιδιαίτερα αυτή στην πρόταση την οποία διατυπώνουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι το δικαίωμα σε ε, δικηγορική αρρωγή να μην ισχύει μόνο για την εκδίδουσα χώρα, αλλά και για τη χώρα εκτέλεσης, ώστε να υπάρχει προστασία και από τις δύο πλευρές της ε, δικαστικής διαδικασίας. Όταν, όταν ε, εκδίδεται ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Η επιπρόσθετη παρατήρηση που θα κάνω σε σύντομη αυτή παρουσίαση είναι και η κύρια ε, ε, διάταξη για τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Είναι σημαντικό βέβαια να υπάρχει πρόσβαση σε δικηγόρο, αλλά αν δεν υπάρχει κάποιο αντιστάθμισμα, τότε τα πράγματα δεν είναι αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε δηλώσεις οι οποίες γίνονται, οι μαρτυρίες οι οποίες συγκεντρώνονται ε, σε περίπτωση παραβίας αυτού του δικαιώματος πρόσβαση σε δικηγόρο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί ε, η καταδίκη ε, ενός ε, υπόπτου, οπότε και παραβιάζουν τα δικαιώματά του. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε αυτή τη διάταξη, η οποία αποθαρρύνει παραβιάσει του δικαιώματος αυτού και που παρέχει την απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Βέβαια, αρχίσαμε να δουλεύουμε με το Κοινοβούλιο και δεί με τον εισηγητή με την έναρξη της ίδιας της πρότασης αυτής και είμαστε ευγνώμονες για τις ανταλλαγές που έχουν λάβει η χώρα. Όπως ξέρετε, η πρώτη ανταλλαγή απόψε έγινε στο Συμβούλιο, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και προσβλέπω στη συζήτηση της πρότασης αυτής μαζί σας. Ευχαριστούμε κυρία Λεμπάη. Και τώρα ανοίγει η συζήτηση για το πρώτο αυτό σημείο ξεκινώντας με την ε, εισηγήτρια, την κυρία Ντονέσκο. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τη Γενική Διευθύντρια για την παρουσίασή τη και ευχαριστώ θερμά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση οδηγία που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί το δικαίωμα σε υπεράσπιση είναι απαραίτητο για μια δίκαιη δίκη. Και αν εξετάσουμε το δικαιικό σύστημα των κρατών μελών, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και όρια σε ό,τι αφορά το δικαίωμα υπεράσπισης. Κάτι που έχει συνέπειες και στην πολιτική της Ένωσης σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση και την εμπιστοσύνη στα δικαιικά συστήματα των κρατών μελών. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι συστάσεις για την Επιτροπή Απαγόρευσης των Βασανιστήριων δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα στα κράτη-μέλη. Και το επίπεδο προστασίας των υπόπτων δεν είναι αρκετό παντού, δεν είναι ε, εφάμιλο παντού. Επίσης χρειαζόμαστε ε, ένα είδος ε, επαγγελματικής νοοτροπίας και μιας κουλτούρας που θα προβλέπει συνδρομή δικηγόρου στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε σχετικά μέτρα. Με την πρόταση αυτή θα σπίζονται κάποια ελάχιστα πρότυπα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των συλληφθέντων ή των υπόπτων σε ποινικέ δίκες, διαδικασίες και το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτον. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τις διατάξεις που αφορούν την εμπιστευτικότητα μεταξύ δικηγόρου και πελάτου. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο εμπιστευτικό χαρακτήρα, ο απόρριτο χαρακτήρα των συζητήσεων μεταξύ του υπόπτου και του δικηγόρου του. Στο απόρριτο αυτό περιλαμβάνονται και οι τηλεφωνικές συνομιλίες και η ανταλλαγή αλληλογραφία μεταξύ δικηγόρου και υπόπτου. Συμφωνώ και με τη διπλή σύσταση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πιστεύω ότι είναι σημαντική η νομική συνδρομή. Χάρη σε αυτή θα λειτουργήσει καλύτερο ο μηχανισμός και θα εξαλειφθούν και κάποιοι μηχανισμοί που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη. Περιμένω τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολλά και διάφορα θέματα. Καταρχήν, ως προς τον στόχο της οδηγίας. Κάποιοι εξέφρασαν ανησυχίες για το γεγονός ότι το ανακριτικό όργανο σε περίπτωση ποινικών διαδικασιών θα πρέπει αυτό ο ανακριτής να εξασφαλίσει τη νομική συνδρομή για τις μικρές παραβάσεις για πτέσματα. Ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του δικηγόρου να εξακριβώσει τις συνθήκες κράτησης. Θα ήθελα κάποιες επεξηγήσεις. Ο δικηγόρος είναι αυτός που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Δίνεται όμως ο δικηγόρος να ελέγξει ή να έχει δικαίωμα ελέγχου των συνθήκων κράτησης του πελάτη του. Έχω και ένα σχόλιο σε σχέση με την ανησυχία που εξέφρασαν κάποια κράτη-μέλη ως προς γεγονός της δυσκολίας εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γίνει αξιολόγηση του κόστους ενσωμάτωσης οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο το κόστος εξαιτίας ε, κάποιων καθυστερήσεων στις ε, διαδικασίες συνεργασίας σε τέτοια θέματα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία και με τους σκιώδεις συγητές. Εγώ ασχολήθηκα και με δύο επιπλέον μέτρα ε, του οδικού χάρτη. Ο κύριος Μπουσουτήλ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επιτροπή για την καλή παρουσίαση της προτάσης αυτή. Αυτή είναι μια πρόταση που δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει μαζί της. Μπορούμε να διαφωνήσουμε με το δικαίωμα ε, του υπόπτου όσον αφορά την πρόσβαση σε δικηγόρο. Και πιστεύω ότι αυτή η πρόταση ε, ε, είναι πολύ σημαντική για μια δίκαιη δίκη και για να διατηρήσουμε και να υποστηρίξουμε την αρχή ότι όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι υποδείξεις του εναντίου. Έτσι, επίσης, από μέρους μου θα ήθελα να εκφράσω την ε, υποστήριξή μου στην πρόταση αυτή. Ε, τώρα, έχω δύο ερωτήσεις για την κυρία Λεμπάη και ελπίζω πως θα είστε σε θέση να τις απαντήσετε. Καταρχάς, κάποια κράτη-μέλη έχουν αντιδράσει σε αυτή την πρόταση λέγοντας ότι εάν πλήρη πρόσβαση στον κατηγορούμενο σε δικηγόρο, αυτό ενδέχεται να παρεμποδίσει τον κατηγορούμενο να πει την αλήθεια, να απαντήσει σε ερωτήσεις και αυτό θα κάνει την, ε, τις έρευνες της αστυνομίας πιο δύσκολες για την ίδια την αστυνομία. Θα ήθελα να έχω την απάντηση της Κομισιόν σε αυτό και πιστεύω πως ε, είναι σημαντικό Κύριε ερώτησή μου. Έπειτα, η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυρία Λεμπάιλ είπε ότι αυτό που κάνουμε εδώ στην ουσία είναι ενσωμάτωση στην νομοθεσία των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισχύει αυτό ή αυτή η πρόταση πάει πέρα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής γνωρίζουν ότι πρέπει να ασκήσουν κριτική στην Κομισιόν όσον αφορά την ε, πρόταση αυτή. Ε, η Κομισιόν χρειάζεται την υποστήριξη και θα την έχει από μας. Πιστεύω όμως ότι εδώ η ερώτηση είναι πολιτική έχει να κάνει με το αν θα διατηρηθούν τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Τα δικαιώματα των κατηγορουμένων από τη μία, τα δικαιώματα του κράτους από την άλλη. Ορισμένα κράτη-μέλη διατύπωσαν ήδη αμφιβολίες. Για κάθε ερώτηση μπορούμε να βρούμε και ένα παράδειγμα για να ε, υποστηρίξουμε ότι αυτό δεν είναι καλό. Επίσης, όμως, υπάρχουν και αρκετά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι είναι βλεβαρό για τους ε, κατηγορουμένους που δεν έχουν δικηγόρο. Πρόσφατα είδα μια αμερικανική αστυνομική ταινία όπου συλλαμβάνεται ο ύποπτο, του διαβάζουν αμέσω τα δικαιώματά του, έχει το δικαίωμα να μείνει σιωπηλό, το δικαίωμα σε δικηγόρο. aber in unseren europäischen Mitgliedstaaten nicht. Αυτός που έχει συλληφθεί είναι μαφιόζος και φυσικά καλεί αμέσως το δικηγόρο του. Πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε, όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και να πούμε ότι το δικαίωμα της νομικής αρρωγής είναι βασικό Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα γιατί θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό το δικαίωμα αυτό. Στη Γερμανία υπήρξαν τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές περιπτώσεις όπου παιδιά απήχθησαν και δολοφονήθηκαν. Ορισμένοι από τους δράστες βρέθηκαν, συλλήφθηκαν. Κάποιοι ύποπτοι ε, συλλήφθηκαν, οι οποίοι όμως δεν ήταν ένοχοι. Είναι σημαντικό ότι Είναι σημαντικό αυτοί οι ύποπτοι να είχαν νομική αρρωγή. Η οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν είναι ε, μόνο μια οδηγία που αφορά δικαστικά ζητήματα, όμως είναι και πολιτική οδηγία. Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και να ενσωματωθεί. και μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λότφορντ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως υπόθηκε, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση. Όταν κάποιος συλλαμβάνεται στο εξωτερικό σε ένα άλλο κρατός μέλος, να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει νομική βοήθεια. Είναι απαραίτητο και καλωσορίζω εγώ και εκ μέρους της ομάδας μου το μέτρο αυτό γιατί φοβάμαι ότι πολλά κράτη-μέλη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το, δικαστή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ομολογία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ε, διεξάγονται ανακρίσεις πριν ο κατηγορούμενος έχει την ευκαιρία να μιλήσει σε δικηγόρο και αυτό είναι απαράδεκτο ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αμοιβαία αναγνώρισης και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ντάλματος Σύλληψης, όπου αναμένεται να υπάρχει συνεργασία. Καλή παρά παραποτέ. Εργαζόμαστε τώρα πάνω στον οδικό χάρτη. Και το σημείο αυτό είναι, όπως είπα, ιδιαίτερα σημαντικό. ιδιαίτερο, ιδιαίτερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχω στην πρόταση ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα σε δικηγόρο στο κράτος που εκδίδει το ένταλμα σύλληψης, καθώς και στο κράτος που εκτελεί το ένταλμα αυτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η νομική σύγχυση και αβεβαιότητα έχει προκαλέσει ε, έχει φέρει δυσάρεστες συνέπειες για τους κατηγορούμενους. Έχουν γίνει εφέσεις επίσης, έχουν γίνει ε, κρατήσεις που δεν ήταν απαραίτητο να γίνουν. Και όλη η διαδικασία αυτή ήταν επίσης και πολύ ακριβή. Γουρά, θα μπορούσε να, διευκολυνθεί η επικοινωνία ανάμεσα στο κράτος που εκδίδει το ένταλμα και στο κράτος που το εκτελεί. Θα μπορούσε η καλύτερη επικοινωνία να αποσύρει μάλιστα και, το, και την εντολή του ένταλματος συλλήψης σε περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος. Εάν, θα μπορούσαν αυτά λοιπόν να είχαν αποφευθεί εάν η πρόσβαση δικηγόρο ήταν δυνατή από την αρχή. Η έκθεση αυτή πρέπει να είναι αξιόπιστη και ρεαλιστική. Όσον αφορά τα, δίκαια, τα, δικαιώματα στις ε, ποινικές διαδικασίες, ελπίζουμε να φέρουν αποτελέσματα. Είμαι απογοητευμένη όμως ότι η χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αποφασίσει να περιμένει μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων για να δει εάν και ελπίζω να το πράξει, διότι εκατοντάδες Βρετανοί πολίτες κάθε χρόνο συλλαμβάνονται σε διαφορετικό κράτος και χρειάζονται ένα τέτοιο μέτρο νομικής αρρωγής. Ωστόσο, όσον αφορά το έγγραφο που συντάχθηκε από πέντε κράτη-μέλη, θα παίξω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ, αλλά κατανοώ κάποιες από τις ερωτήσεις που έχουν προκύψει. Για παράδειγμα, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λεμπέλ στην πρόταση της Επιτροπής. Στα σχόλια για το άρθρο 4, για το περιεχόμενο του δικαιώματος πρόσβασης στο δικηγόρο. Το σχόλιο λέει ότι η πρόταση έχει ως εξής ότι παρουσία Η παρουσία δικηγόρου είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε διαδικασία συγκέντρωση ή παρουσίαση αποδείξεων. Στην υπόθεση Τάνεν εναντίον Τουρκίας, όπως ε, θα δείτε, το κοίταξα χθε, έχει να κάνει ε, αποκλειστικά με την σύλληψη από την αστυνομία, με την κράτηση από την αστυνομία. Όλες οι υποθέσεις που αναφέρονται έχουν να κάνουν με τη στέρηση ελευθεριών και την ε, αστυνομική κράτηση. Ποια είναι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την παρουσία δικηγόρου στην συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Στα πλαίσια της ε, προδικασίας. Πόση ουσία πραγματικά υπάρχει σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να παρεμποδιστεί η διαδικασία συλλογής αποδεκτικών στοιχείων, ότι ο δικηγόρος ε, χρειάζεται, εάν κάποιο, για παράδειγμα συλληφθεί στον δρόμο επειδή οδηγεί μεθυσμένος ή στη διαδικασία λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πιστεύω ότι χρειάζεται, χρειάζονται περισσότερε εξηγήσει αυτό. Επίσης ελπίζω να συζητήσουμε το κόστος που θα εμπίπτει. Πιστεύω πως, όπως είπα και πριν, η επένδυση στη δικαιοσύνη μπορεί να μας ε, εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Όσον αφορά τώρα κάτι άλλο, η πρόσβαση σε, τηλέφων, σε τηλεφωνική επικοινωνία θα αποκλειστεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Τέλος, θα έπρεπε αυτή η πρόταση να συντάξει κανόνες σχετικά με το την παραδεκτότητα των αποδεκτικών στοιχείων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω τα κράτη-μέλη... Κύριε Άλμπρεχτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Δεν είμαι μόνο σιώδης για την ομάδα μου, αλλά και η συγητής της ε, Γνωμοδότης Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων στο θέμα αυτό. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έλαβε χώρα χθε στη συνάντηση Γιούρη και είχαμε μια συνάντηση με τους σκιώδους ηγητές στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προσπαθώντας να γνωμοδοτήσουμε το συντομότερο δυνατόν ώστε να συμπεριληφθεί η άποψή μα και στη διαδικασία στην εδώ Επιτροπή. Και θα ήθελα να ζητήσω από όλους μας να σεβαστούμε την άποψη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, θέλει να παρέμβει, και να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε την άποψη της στην έκθεσή μας. Όντας όμως και όδη και για την ομάδα μου, θα το φροντίσω. Νομίζω, όπως ε, ήδη επισημάνθηκε από τους άλλους και ηγητές των άλλων ομάδων, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικός φάκελος και ως βουλευτές πάντα ζητούσαμε αυτό τον οδικό χάρτη όπου αναδύεται αυτό το μέτρο για την ε, ύπαρξη δικηγόρου σε όλες τις ποινικέ ε, διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την κίνηση αυτή και ιδιαίτερα διότι είχαμε χρόνια ε, θέσπισης μέτρων αμοιβαίας αναγνώρισης, όπου υπήρξαν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις όπου τα ατομικά δικαιώματα και δικαιώματα υπόπτων δεν θεωρήθηκαν ένα θέμα στο οποίο χρειαζόταν εναρμόνιση των ε, νομικών ε, συστημάτων και ότι χρειαζόταν να έχουμε ενιαίες προδιαγραφές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως τώρα βρίσκεται διαδικασία, με τη διαδικασία συναπόφασης μετά τη συνθήκη της Λισαβόνα θέλει να θεσπίσει αυτά τις ελάχιστες προδιαγραφές. Και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι βέβαια πολύ ψηλό επίπεδο ελάχιστων προδιαγραφών για τα δικαιώματα των ατόμων. Και όχι μόνο το ελάχιστο, το μήνυμο μινιμόρουμ το οποίο υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι νομίζω και ο λόγος για τον οποίο υποβάλλουμε αυτή την πρόταση. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει, όπως είπε η κυρία Ζήπε, να διασφαλίσουμε τα υψηλά επίπεδα ατομικών και διαδικαστικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ε, ευθυγραμμιστούμε στην βάση όταν συνεργαζόμαστε για θέματα αστυνομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό για πάρα πολλά κράτη-μέλη αυτό το διάβημα. Έχω κάπως την εντύπωση ότι κάποια από τα κράτη-μέλη τα οποία τώρα πιέζουν ε, πατάνε το φρένο, ενώ θα έπρεπε να επιταχύνουμε στην εισαγωγή κοινών προδιαγραφών, είναι αυτοί που από την άλλη πιέζουν για μεγαλύτερη συνεργασία σε θέματα αστυνόμευσης και δικαιοσύνης. Σκέφτομαι για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκή Εντολή ε, Ερευνών, είναι το πεδίο όπου όλε οι κυβερνήσει των κρατών μελών λίγο πολύ συμφωνούν, ιδιαίτερα χώρε όπω το Βέλγιο και η Γαλλία. Εκεί θα περιμένω ότι θα κατανοούσαν ότι η μεγαλύτερη συνεργασία και περισσότερη αμοιβαία αναγνώριση μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν έχουμε ταυτόχρονα και ελάχιστε προδιαγραφέ για ποινικέ ε, κυρώσει και διαδικασίε και σε ό,τι αφορά την προστασία ατομικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι όλοι μας και σε όλες τις πολιτικές ομάδες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο θα το υποστηρίξουμε και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία όταν θα συντάσσουμε την έκθεσή μας πάνω στο θέμα αυτό. Ως εκ τούτου υποστηρίζω την εργασία του εισηγητή και θα συνεργαστώ στενά μαζί του, υποστηρίζοντας τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής και επιλύοντας το ανοιχτό ερώτημα που βρίσκεται επιτάπητος. Νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Αρκεί να αναφέρω ένα μόνο. στο ζήτημα παρουσίας δικηγόρου όταν συλλέγονται πιστήρια ή όταν ε, διεξάγονται έρευνες στην όλη διαδικασία, όταν κάποιος είναι ήδη ύποπτος σε μια ποινική ε, δίωξη, Μπορεί να υπάρξουν βέβαια εξαιρέσει όπου θα απαγορεύεται να είναι παρόν συνήγορο κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να μην επιτρέπεται να είναι παρόν κάτι διάρκεια διεξαγωγή, προτού ολοκληρωθεί κάποια έρευνα. Θα πρέπει να υπάρχει όμως η αρχή ότι ένας ύποπτος σε ποινική, ε, που υπόκειται σε ποινική δίωξη θα πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβαση σε συνήγορο και να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τα δικαίωμά του σε όλες τις φάσεις και τις διαδικασίες, σε όλες τις φάσεις διαδικασίας. Γιατί χωρίς, αν δεν τα γνωρίζει τα δικαιώματά του στι ε, διαδικασία αυτή, κανεί δεν μπορεί να φροντίσει και να προασπίσει τα δικαιώματα αυτά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσει σε κράτη-μέλη όπου οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση των δικαιωμάτων του και γι' αυτό ακριβώ δεν μπορούν προφανέστατα και να τα χρησιμοποιήσουν και να τα επικαλεστούν κατά τη διάρκεια ποινικών διώξεων. Ο κύριος Κίρκοπ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όταν βλέπει κανείς μια ωραία τούρτα του φαίνεται καλά αρεστή μέχρι που παίρνει το μαχαίρι και την κόβει και διαπιστώνει την πραγματική της ουσία. Φυσικά όλα φαίνονται σαν ωραίο κέικ μέχρι στιγμής, πολύ δύσκολα κανείς θα διαφωνούσε. Αλλά πολύ σωστά επισήμαναν οι προλαλήσαντες ότι χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια και φυσικά Ενάργεια ως προς τους ορισμούς. Καταρχήν να είμαστε σαφείς ως προς το τι, ποιος είναι δικηγόρος, με ποιο τρόπο κανείς μπορεί να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο. Δεν μιλούμε για ε, πληρεξούσιο δικηγόρο. Επίσης, τι είδους πρόσβαση εννοούμε. Άμεση πρόσβαση, τηλεφωνική πρόσβαση, το τηλέφωνο περιλαμβάνεται, όπως επισήμανε η κυρία Λάντφορτ. Όλα αυτά είναι σημαντικά να τα διευκρινίσουμε σε πολλές... Ε, σε πολλά δικαιϊκά συστήματα αρκεί πρόσβαση σε τηλέφωνο. Ε, το τηλέφωνο στο δικηγόρο θεωρείται αρκετή εγγύηση. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει μια συνολική πρόταση, καλύπτοντα όλα τα δικαιώματα υπεράσπιση σε ποινικέ δίκε, ακόμη και τέτοια ζητήματα, αλλά ουδέποτε δεν εγκρίθηκε η πρόταση αυτή από το Συμβούλιο για τον απλούστατο λόγο ότι όταν κάποιο ε, ασχολείται με οικουμενικά ελάχιστα πρότυπα, είναι πολύ δύσκολο με τόσο διαφορετικά δικαιϊκά συστήματα και διαφορετικές δικονομίες να εφαρμόσουμε έστω και ελάχιστα πρότυπα. Και το θέμα του κατά πόσο και πότε ένας ε, δικηγόρος έχει επαφή και όχι μόνο το είδος της επαφής είναι σημαντικό. Και το αργότερο κατά τη στέρηση της ελευθερίας. Και αυτό το θέμα όμως ε, χρήζει διευκρίνησης. Πότε θεωρείται κάποιος ότι στερείται της ελευθερίας του θεωρείται στέρηση ελευθερίας η κράτηση η σύλληψη στο δρόμο ή θεωρείται στέρηση ελευθερίας μόνο εφόσον κάποιος ε, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα ή μεταφέρεται στο κρατητήριο. Πότε ξεκινάει η στέρηση ελευθερίας και αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Και κάτι άλλο, επιπλέον πόροι που απαιτούνται δεν εξετάστηκαν αρκετά διεξοδικά. Για παράδειγμα δεν έχουμε μελέτη επιπτώσεων οικονομικών, ούτε αντιλαμβανόμαστε την πολυσύνθετη φύση αυτής της νομικής συνδρομής και το σύστημα προβών που υπάρχει σε πολλές δικαιοδοσίες. Βέβαια, καλό είναι να έχει κανείς δωρεάν νομική συνδρομή, αλλά όταν έχουμε νομική συνδρομή και υπάρχει κόστος σε πολύ πρόημο στάδιο από αυτό που προτείνεται, σε οποιαδήποτε διαδικασία κάποιος θα πρέπει να λάβει τα έξοδα και αυτά να τα διευκρινίσουμε θα ήθελα αν προχωρήσουμε και εγκρίνουμε την πρόταση, δεν την επικρίνω. Είναι δικαίωμα πρόσβαση ε, σε δικηγόρο κατηχερωμένο και, και εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν θέλω να στερήσω από το, από το επάγγελμά μου τη δυνατότητα να έχουν επαφή με υπόπτου οι πελάτε. Αλλά προσοχή, πριν από μια επταετία δεν καταφέραμε να εγκρίνουμε την αντίστοιχη πρόταση. Το Συμβούλιο επισήμανε επιφυλάξει και ανησυχίε. Το ίδιο και τώρα για πολλούς ε, λόγους που σας εξέθεσα πριν από λίγο. Οπότε, είμαι υπέρ, υπό όρους όμως, και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει σαφείς ορισμούς για τα ζητήματα που ανέφερα και εγώ αλλά και άλλοι, αν λάβουμε αυτές τις διευκρινήσεις, νομίζω ότι θα είμαστε πιο ικανοποιημένοι με την πρόταση. Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω ογκρικά. Előtt, még valószínűleg furcsán néztek volna, vagy haragudtak volna. Θα ήθελα να... Ε, να ε, υπερασπίσουμε ακριβώς αυτή, αυτή την πρόταση προστασίας ε, των ε, υπόπτων ή των κατηγορουμένων. Με, μπορεί κάποιοι να με κοιτάξουν στραβά θεωρώντα ότι θέλω να, υποσ... Ε, εξασφαλίσω δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο από πολύ πρόωρο στάδιο σε υπόπτου. Αυτό δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, το 2002 για παράδειγμα, αλλά στο μεταξύ η Ουγγαρία ε, έχει περάσει από πολλά στάδια και παρόλο ότι στο παρελθόν είχε διαπράξει σημαντικές παραβιάσεις και έχει κάνει μεγάλο δρόμο και μπορεί στην Ουγγαρία με κοίταζε στραβά πριν από μερικά χρόνια μια τέτοια πρόταση. Σήμερα πολλοί μπορούν να συμφωνήσουν. Και πολλοί στην Ουγγαρία διαπίστωσαν τι σημαίνει να στερείται κανείς δικαιώματα και να στερείται ε, εγγυήσεων και δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όταν ε, εμπλέκεται σε μια τέτοια ποινική διαδικασία. Είχαμε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2006, έγινε μια αντικυβερνητική διαδήλωση και πολλοί διαδηλωτές ε, ε, ξυλο, ξυλοφορτώθηκαν, σύρθηκαν στην αστυνομία, κακοποιήθηκαν, ε, υπέστησαν μετά ανάκριση, τους απεγγέλθηκαν διάφορες κατηγορίες και μία από τις υποθέσεις αυτές δημοσιεύθηκε και είχε μεγάλη απήχηση. Επρόκειτο για ένα φοιτητή που είπε σε έναν αστυνομικό που τον ανέκρινε ότι, ε, ότι θα ήθελε νομική συνδρομή, θα ήθελε παρουσία δικηγόρου. Και ο αστυνόμος απάντησε στο φοιτητή ανόητε, ηλίθιε μάλλον. Δεν είμαστε Ηνωμένε Πολιτείε εδώ, δεν έχεις δικαίωμα σε δικηγόρο. Τώρα, ακόμη και στην Ουγγαρία, αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται κανεί νομική συνδρομή, παρουσία δικηγόρου το συντομότερο δυνατό και είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε διάφορε δικονομικέ εγγύησει. Έχουμε διανύσει σημαντικό δρόμο στην Ουγγαρία. Βέβαια, άλλο τα δικαιώματα των αθών και άλλο τα δικαιώματα των ε, ενόχων. Και στην Ουγγαρία το 2002 θεωρούσαμε ότι μόνο οι αθώοι δικαιούνται ορισμένα πράγματα και όχι ένοχοι. Αλλά πολλά άλλαξαν έκτοτε όπως σας είπα και έχουμε και το τεκμήριο της αθωότητας πριν την έκδοση δικαστικής απόφασης. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης, μέχρι την καταδίκη, ο ύποπτο τεκμέρεται αθώος. Οπότε έχει τα ίδια δικαιώματα, άσχετα με το αν θα καταδικαστεί τελικά ή όχι. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αθώου και ενόχου. Όλοι λοιπόν έχουν δικαίωμα σε πρόσβαση σε δικηγόρο, όλοι δικαιούνται δικονομικές εγγύσεις. Nos, τελικά δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει. Πάντως σήμερα βρισκόμαστε σε μία φάση που ακόμη και η Ουγγαρία είναι όριμη να εξετάσει τέτοιου είδους ε, προτάσεις. Έχω μερικές ε, συστάσεις και εγώ κυρία Λεμπάγη. Όπως είπατε, θα πρέπει κανείς σε πρώιμο στάδιο να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο, να τη χάνει νομικής συνδρομής. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι πραγματικά κατεπίγουσες. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το γκρικό δίκαιο δέχεται την αποποίηση αυτού του δικαιώματος ε, νομικής συνδρομής. Εκκινώντας λοιπόν από αυτή την εμπειρία, θεωρώ ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να τεκμηριώσουν την κατεπίγουσα περίπτωση και την α, ε, ολιγορία στην παρουσία του δικηγόρου. Θα πρέπει να γίνει μια αντιστροφή του βάρους απόδειξης και θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να αποδεικνύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με εξαιρέσεις ότι ε, συνέτρεχε κατεπίγουσα περίπτωση και γι' αυτό δεν μπόρεσε να παρίσταται ο δικηγόρος από την προ... πρόορη φάση της διαδικασίας. Κάτι άλλο που θα ήθελα επίσης να επισημάνω. Γνωρίζουμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα σε ποιοτική νομική συνδρομή. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα της ποιότητας. Δικαιούται μια ποιοτική νομική συνδρομή ο πολίτης. Η κυρία Λεμπάι μίλησε και για τις, τη φάση της ε, έρευνας ή της ανάκρισης ε, ή τη συγκέντρωση των αποδείξεων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση έρευνας, είχαμε την περίπτωση τώρα στην Ουγγαρία και είχαμε τέτοιες έρευνες. Ακόμη και σε αυτό το στάδιο της έρευνας χρειάζονται κάποιες οικονομικές εγγύησεις και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Φως. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία κυρία Αντώνεσκου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 2, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σε αυτό. Στην ε, εκδοχή που έχουμε τώρα, τι γίνεται όσον αφορά την ανάκριση, το ένταλμα, πώς θα γίνει η αξιολόγηση των, ε, των ανακρίσεων έπειτα. για μας, για τη Γερμανία, είναι αυτονόητη η άμεση, όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαφή του κατηγορούμενου με δικηγόρο. Στο γερμανικό κείμενο η οδηγία αυτή ονομάζεται το δικαίωμα σε νομική αρρωγή. Στο αγγλικό κείμενο λέμε, βλέπουμε right of access to a lawyer, δικαίωμα σε πρόσβαση σε δικηγόρο. Εδώ θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν να γραφεί και κάτι αντίστοιχο στο γερμανικό κείμενο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία αυτή, που είναι σημαντική, που συνενώνει δύο άλλες οδηγίες, όχι μόνο το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, αλλά και την ε, ενημέρωση ή επαφή με την προξενική αρχή ή τα μέλη της οικογένειας. Πρόκειται για δύο οδηγίε που εκκρεμούσαν πολύ πριν και τη Σουηδική Προεδρία. Η Σουηδική Προεδρία καθόρισε έναν οδικό χάρτη, ένα φύλλο πορεία για αυτό το πακέτο και ευτυχώ, κάλλιο αργά παρά ποτέ, ξεφύγαμε από το αδιέξοδο και καταφέραμε τελικά να προχωρήσουμε σε, αυτή σε αυτό το πακέτο των δύο οδηγιών. Γιατί έτσι φροντίζουμε τουλάχιστον κάποια ελάχιστα πρότυπα να εξασφαλιστούν και κυρίως για τα ευάλωτα άτομα. Και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική προστασία των ευάλωτων ατόμων σε αυτό το δικονομικό πακέτο. Θα ήθελα να υποβάλω και εγώ κάποιες προτάσεις που ήδη διατυπώθηκαν, ερωτήσεις ως προς το πότε ξεκινά αυτό το δικαίωμα γιατί είναι σαφές από το κείμενο ότι στις ανακρίσεις, στην ανακριτική διαδικασία απαιτείται παρουσία δικηγόρου. Είπαμε όμως ότι από τις πρώτες δηλώσεις, οι πρώτες δηλώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδείξεις εις βάρος του υπόπτου. Οπότε ήδη από τη φάση αυτή των αποδείξεων ίσως θα χρειαζόταν παρουσία του δικηγόρου. Στην πρώτη οδηγία που ήμουνα και σκιώδη συγγήτρια για το δικαίωμα μετάφραση και διερμηνίας, και εκεί επιμείναμε στην ανάγκη προσδιορισμού της στιγμής γέννησης του δικαίου. Γιατί και στην στιγμή ε, μετάφραση διερμηνίας επιμείναμε στο πότε γεννάται αυτό το δικαίωμα. Το ίδιο και στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να δούμε πότε ξεκινάει αυτό το δικαίωμα. Γιατί υπάρχουν όντως διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αλλά καλό θα ήταν να δημιουργηθεί μία σύγκληση. Να δούμε Οπότε ο ύποπτο ενημερώνεται για το ότι είναι ύποπτο. Και οι λόγοι για τον εξαιρετικό χαρακτήρα. Αυτοί οι λόγοι παρά ελαστικοί και ανοιχτοί και αφήνουν μεγάλη διακριτική ευχαίρεια στον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας. Γιατί είναι τόσο γενική αυτή η διάταξη. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να διευκρινιστεί περαιτέρω και να περιοριστεί κάπως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε... Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Λεμπάη για την παρουσίασή σας, την εξαιρετικά συνεκτική και σαφή. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία στα, στα σχόλια, τα πολύ άριθμα άλλωστε σχόλια των συναδέλφων που ετέθησαν σε όλα αυτά τα ζητήματα που βέβαια αφορούν σε ένα κείμενο που είναι εξαιρετικά τεχνική υφή, αλλά που είναι θεμελιώδης και βέβαια αρμοδιότητα όχι μόνο της Επιτροπής μας, αλλά και άμεσα πηχώντας ε, το κατόφλι των ευρωπαϊκών ιδεών και αξιών που απηχούμε. Και η όλη συζήτηση ουσιαστικά αποδεικνύει πόσο κοινή είναι αυτή η πλατφόρμα για όλους μας και τα ζητήματα και τα ερωτήματα οποία σε τέθησαν είναι ακριβώς διευκρινιστικά, είναι ορισμών, είναι ε, καθορισμού παρά ουσίας σε ό,τι αφορά τα θέματα ατομικών ελευθεριών που είναι δύσκολο να παρακολουθεί στα πλαίσια δημιουργίας μιας ενιαίας Ευρώπης δικαιοσύνης όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη συζήτηση μεταξύ των κρατών, γιατί όλοι έχουμε, αν θέλετε, εγκαλιστεί από τις διαφορετικές θέσεις των κρατών μελών, αλλά και που αφορούν στο καθεστώς του Ευρωπαίου πολίτη. Δηλαδή το ενδυνάμει δικάσιμο που μπορούμε να είμαστε και το ενδυνάμει των θυμάτων που μπορούμε να είμαστε όλοι. Αυτή η δύσκολη σε ψεφίτευξη ισορροπία πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του τεκμηρίου αθεότητας και εξασφάλισης του θεμελιώδους δικαιώματος υπεράσπισης που θέλει να δημιουργήσει το κείμενο αυτό και ο σεβασμός του ο κανόνας του σεβασμού των δικαιωμάτων και η κύρωση εφόσον υπάρχει παραβίωση των δικαιωμάτων αυτών και ακριβώς η αναγκαιότητα ε, διεξαγωγής ε, ερευνών προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Η συλλογή αποδείξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικές και διαυγείς. Χωρίς να μακρηγορώ λοιπόν και χωρίς να ε, επιμένω σε κάποια ερωτήματα τα οποία θα απαντήσετε και που με ενδιαφέρουν, θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω την προσοχή σας σε κάποιους ε, ορισμούς και κάποιες ε, αποσαφηνίσεις σε ό,τι αφορά τις πιθανές παρεκκλήσεις σε ό,τι αφορά την παρουσία συνηγόρου. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω ποια είναι η θέση σας σε ό,τι αφορά την πραγματική δικαστική αρρωγή. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα θέματα κόστους, αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, όλη διαδικασία. Αν θέλουμε να είμαστε πλήρεις, νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό, ώστε να επιτρέπεται στα άτομα που ίσως βρίσκονται σε χρηματική δυσκολία, να μπορούν να απολαμβάνουν του ιδίου των δικαιωμάτων όπως και οι άλλοι είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί πραγματικά να ανταπαντήσει σε κάποια ερωτήματα και να κάνει πολύ πιο στιβαρό το κείμενο αυτό. Θα ήθελα επίσης να θέσω ερωτήματα πάνω στην πρόταση που γίνεται στο σημαντικό αυτό κείμενο, να, ζητηθεί, ζητείτε από τους ε, να διεξάγουν κάποια έρευνα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης ενός υπόπτου. Προφανώς και πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Και μάλιστα η χώρα μου δεν είναι μεταξύ των πλέον ε, ικανοποιητικών και αποτελεσματικών σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά είναι αρμοδιότητα των συνηγόρων να κάνουν τέτοιου είδου έρευνα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δώσει κάποιες σχετικές απαντήσεις. Υπήρχε και ένα ερώτημα ουσίας το οποίο είχα ξεχάσει. Ε, την πολύ καλή διατύπωση ε, ε, που είπε η παρακαθήμενη ότι θα παίξει το ρόλο, του δικηγόρου του διαβόλου. Και εγώ αντίστοιχα θα επιθυμούσα ή δυνατόν να μας απαντήσετε σε αυτή την αντίρρηση παρουσία συνηγόρου από την πρώτη στιγμή κράτησης. Πράγμα το οποίο μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι η παρουσία συνηγόρου ίσως επιβραδύνει τη συλλογή στοιχείων. Ευχαριστούμε. Ο εκπρόσωπος της ε, Πολικής Προεδρίας, Πολωνικής Προεδρίας, ίσως θα πάρει το λόγο, πρωτού δώσουμε και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για αυτή την πρόταση. Πολωνική Προεδρία εργάζεται στο Συμβούλιο για, πάνω σε αυτό το κείμενο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο δικός χάρτης της Κομισιόν και των... ήταν δέσμευση των κρατών μελών να επεξεργαστούν τα μέτρα που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή. Ήδη τονίστηκε από πολλούς ομιλητές ότι είναι από τα σημαντικότερα μέτρα και από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά τους κατηγορούμενους και το δικαίωμά τους πρόσβασης σε δικηγόρο. Πιστεύω πως όλοι το συμμεριζόμαστε αυτό. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο το εξετάζει προσεκτικά. Ήδη είχαμε την πρώτη συζήτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών και το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει από αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τα μέτρα αυτά. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα που πρέπει να ε, διαλευκανθούν όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής. Από, από τη σκοπιά των κρατών μελών τώρα, όταν, ε, εάν δούμε τη θέσπιση προτύπων, θα δούμε πως είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη κάποια στοιχεία που βρίσκονται στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα κράτη-μέλη όταν επεξεργάζονται οποιαδήποτε νομοθεσία. Η νομολογία του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πάντα τονίζει την ποιότητα. Από τη μία έχει να κάνει με το να δίνει δικαιώματα δικής δίκης στον κατηγορούμενο, από την άλλη επιτρέπει στις αρχές να διεξάγουν μία αποτελεσματική ποινική διαδικασία. Και αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Γιατί αυτή η πρόταση έχει να κάνει με τα κοινά ελάχιστα πρότυπα στις ποινικέ διαδικασίες. Κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν εδώ ε, μίλησαν για εξειδικευμένες αναλύσεις. Γιατί το αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στην ουσία στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη-μέλη είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε υπόψη. Πρέπει να, να, έχουμε υπόψη τον στόχο. Ο στόχος είναι η δικαιοσύνη στα θύματα Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι όπως αναφέρθηκε, η, μια δικαιοσύνη που καθυστερεί είναι μια δικαιοσύνη που δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναλύσουμε ε, διεξοδικά το αντίκτυπο της πρότασης αυτής. Και επίσης να αναλύσουμε το κόστος και τον τρόπο εφαρμογής κάποια από τα μέλη ήδη τόνισαν ε, ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα νομικά συστήματα της κάθε χώρας και ότι είναι δύσκολο να βρεθούν κοινά πρότυπα που θα γίνουν αποδεκτά από όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή διεξάγουμε αναλύσεις πάνω στην, πρόταση αυτή, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και ενυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας πάνω σε αυτό και ελπίζουμε σε καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με την Κομισιόν πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Λεμπάη. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη μου αντίδραση είναι ότι πραγματικά ενθαρρύνομαι ιδιαίτερα από τη συνολική υποστήριξη που εκφράσατε σήμερα για την πρόταση αυτή όπως είπα και προηγουμένως, είναι η πλέον σημαντική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πλέον σημαντική από όλα τα διαδικαστικά δικαιώματα τα οποία έχουμε προτάξει μέχρι στιγμής. Νομίζω, προτού έρθω να απαντήσω στα ερωτήματά σας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν το 2004. Γιατί εντωμεταξύ είχαμε την υπόθεση Σαλντούς και είναι υποστή υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη να μην ε, υποπέσουν κάτω από αυτά που μας δίδαξε αυτή η υπόθεση. Προσπαθήσω όμως τώρα να απαντήσω τα ερωτήματά σας. Και θα απαντήσω με τη σειρά των παρεμβάσεων. Ξεκινώ με την εισηγήτρια λοιπόν, την κυρία Τουντέσκου. Θέσατε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το ε, μικρό, μικρό παράπτωμα. Ήταν ερώτημα που ανέφερε και η Σάρα Λότφορντ όταν αναφέρθηκε στο άρθρο 4. Εάν δηλαδή κάποιος, θα σταματήσει κάποιος στην άκρη του δρόμου για να ε, κάνετε το τεστ, το αλκοτέστ, έχετε δικαίωμα να πείτε δεν πρόκειται να φυσήξω αν δεν έχω παρουσία δικηγόρο. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το, θέλω να το κάνω σαφέ, όπω το έκανε και ο Αντιπρόεδρο κατά τη διάρκεια τη συνάντηση του Συμβουλίου, όταν είπε ότι για την λήψη δαχτυλικών αποτεμάτων ή για αλκοτέστ ή για τέτοιου είδου ε, παραπτώματα ή μικρή ε, ε, μικρής σημασίας ε, πράξης, προφανώς δεν πρόκειται να παρακολύσουμε την όλη διαδικασία να την επιβραδύνουμε με την επιβολή Τη υποχρέωση παρουσία συνηγόρου. Αυτό το θέμα λοιπόν παρουσία συνηγόρου εν πολλής προσπαθεί να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ τη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πάντων, συμπεριλαμβανομένων και των υπόπτων και εξασφάλιση του ότι οι περιπτώσεις αυτές και οι διώξει θα μπορούν να προχωρούν και να μην επιβραδύνεται η όλη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Νομίζω ότι ζητήσατε επίσης ε, ρωτήσατε και περί της όλων αυτών των μέτρων και του κόστους που, που συνεπάγεται. Το πρώτο που θέλω να πω ότι είναι ότι υπάρχει σειρά κρατών μελών που έχουν ήδη μεταφράσει την πρόταση αυτή και μεταφέρει σε εθνική νομοθεσία. Και βέβαια σε διαφορετικές φάσεις το κάστος ίσως στην αρχή μπορεί να είναι λίγο υψηλότερο. Αυτό ισχύει και για τα θέματα ε, δικηγορικής ε, αρρωγής που έθεσαν αρκετά μέλη του, Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, θα σχολιάσουμε σχετικά με αυτό στη συνέχεια, δεν μας ευχαριστεί να υπάρξει επιβάρυνση του κόστους, όμως εάν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και προτού υιοθετηθεί το θέμα ε, αρρωγής δικαστικής, ε, αρρωγής ε, υπεράσπισης, ουσιαστικά θα ισχύει και θα κυριαρχεί η εθνική νομοθεσία έναντι της κοινοτική. Έρχομαι στο ερώτημα του κ. Βουζουτήλ που ουσιαστικά μας λέει το εξή. Δεν θεωρείτε ότι η παρουσία δικηγόρου ίσως εμποδίσει ή αν θέλετε αποτρέψει τον ύποπτο από το να πει εξ αρχή την αλήθεια και είναι μία από τις ανησυχίες που εκφράζουν κράτη-μέλη. Νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα αυτό με διαφορετικό τρόπο. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, σε μια σειρά περιστάσεων τότε, άνθρωποι που είναι απόλυτα αθώοι, οδηγούνται στο να αποδεχθούν ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα, γιατί αισθάνονται χαμένοι στην όλη διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ότι στην περίπτωση των ατόμων εκείνων που ε, είναι ύποπτοι, αλλά αποδεικνύεται ότι περίτραναν στο τέλος της διαδικασίας ότι είναι αθώοι, και δεν έχουν διαπράξει καμία παραβίαση του νόμου για την οποία, για την ήταν ύποπτη στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς την περιπτώση λοιπόν υπάρχει συνήγορος. Εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται κάποιος ε, κατηγορούμενος από την αλήθεια. Αν δηλαδή υπάρχει παρουσία συνηγόρου μπορούμε να τον συμβουλεύσουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποτραπούν οι δυνάμεις καταστολής, οι δυνάμεις του νόμου δηλαδή, από το να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ανάκριση του υπόπτου. Τώρα και σε ό,τι αφορά το ερώτημα του ε, αν μπορούμε να υπερβούμε αυτό που μας λέει η δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην περίπτωση στην υπόθεση Σαλντούς, δύο σχόλια έχω να κάνω. Καταρχάς θα έλεγα ότι αυτό που κατά βάση κάνουμε είναι να μεταφράζουμε στην πρόταση αυτή την δικαστική απόφαση του δικαστηρίου. Υπάρχουν βέβαια αποκλήσεις σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και είναι εξίσου αληθές ότι στην πρόταση αυτή έχουμε υιοθετήσει μια ερμηνεία η οποία είναι ευνοϊκή προς τον κατηγορούμενο. Δεν το αρνούμαστε. Όμως πιστεύουμε ότι εξίσου, επειδή ακριβώς πιστεύουμε έντονα ότι η πρότασή μας δεν μπορεί να βρεθεί κάτω από τον πύχη της ε, δικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι είναι λοιπόν τα σημεία στα οποία ξεπερνούμε αυτό το οποίο μας είπε το δικαστήριο. Το ένα είναι στο δικαίωμα επικοινωνία, το οποίο δεν είχε εξασφαλιστεί στην υπόθεση Σαλτούς, αλλά το οποίο είναι ένα θεμητό δικαίωμα των ε, ανθρώπων όταν είναι ύποπτοι να μπορούν να πούν στον εργοδότη, στους οικείους τους, ότι είναι σε κράτηση, είναι ύποπτοι και να εξηγούν γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν αυτό δεν επιτρέπεται σε πολλά κράτη-μέλη και το άλλο στοιχείο το οποίο επισημαίνω εδώ είναι η περίπτωση που αναφέρθηκε και πάλι από τη Σάρα Λάτφορντ και που είναι το δικαίωμα σε δικηγόρο σε περίπτωση ευρωπαϊκής νομολογίας στην εκδίδουσα χώρα. Πράγμα που στο παρόν δεν ισχύει. Αυτές είναι ουσιαστικά οι δύο διατάξεις που δεν είχαν ουσιαστικά συζητηθεί στην ε, υπόθεση Σαλντούς. Τώρα, πάνω στα θέματα διευκρίνησης που απαιτούνται και απαντώ με αυτό στο ερώτημα που έθεσε κ. Κίχοφ. Το ζήτημα δηλαδή του τι είδους πρόσβαση σε δικηγόρο επιθυμούμε. Θα λέω και πάλι ότι αυτά είναι πράγματα που πρέπει να διευκρινίσουμε όταν αναφέρουμε πρόσβαση εννοούμε φυσική την παρουσία ή τηλεφωνικά. Θα είναι αντικείμενο συζήτηση που θα έχουμε και μαζί σας και με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε. Η κυρία Σμουβά έθεσε το ερώτημα της παράκαμψης, δηλαδή τι συμβαίνει εάν το δικαίωμα αυτό δεν γίνεται σεβαστό. Είπαμε λοιπόν ότι το κράτος θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν ισχύει γιατί τι σημαίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι σεβαστό ο νόμος αυτός. Νομίζω ότι πάμε και παραπέρα. Δείτε το άρθρο 17 της οδηγίας αυτής. Αναφέρεται ότι η διακήρυξη που θα γινόταν χωρίς την παρουσία δικηγόρου δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το σκεφτούμε καν. Προτού το κάνετε λοιπόν, ουσιαστικά αφαιρείται από κάποιον το δικαίωμα σε συνήγορο. Πρέπει να σκεφτείτε τις συνθήκες αυτές και το πρόβλημα ιδιαίτερα που σας δημιουργεί. Θα κληθείτε σε ανάκριση. Νομίζω λοιπόν ότι στο άρθρο 13 έχουμε σχεδιάσει αυτό το προηγούμενο. Στο άρθρο 12, κύριε θα το κοιτάξουμε. Ε, αναφέρεται ο τίτλος στα γερμανικά. Θα το εξετάσουμε και αυτό. Και τώρα ε, στρεφόμενοι στην κυρία Ρομέρο. Θέσατε δύο ερωτήματα. Το πρώτο, πότε θα καταλήξουμε σε μια λογική απόφαση. Σκοπεύουμε να έχουμε ολοκληρώσει μια πρόταση μέχρι του χρόνου. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη και, τους, ε, ε, και τον πληθυσμό Ρωμά, Συγγνώμη για τους πλέον ευάλωτους, γιατί η πρότασή μας ε, ισχύει για όλους όσοι είναι υπόπτοι. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές χώρες μέλη η έννοια του υπόπτου δεν υφίσταται αυτή υπαρκτή. Γνωρίζουμε ότι είσαι ύποπτος όταν αρχίζουν να εμφανίζονται και να συλλέγονται στοιχεία, οι μαρτυρίες που συνηγορούν, αν θέλετε, και που επιβαρύνουν την κατάσταση στην διάπραξη ή συμμετοχή κάποιας παράβασης. Όμως, στο θέμα της, ε, στη διαδικασία της ανάκρισης, μιας πρώτης ανάκρισης του πότε θεωρείσαι ύποπτος, είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι ένα θεμητό ερώτημα και το έχουν θέσει πολλές, ε, πολλά κράτη-μέλη. Κυρία Γκρίσμπεκ, θα σας απαντήσω στα γαλλικά θέτεται το ερώτημα της ε, νομικής αρρωγής και νομίζω ότι εν μέρει έχω απαντήσει το ζήτημα αυτό. Θα επανέλθουμε δηλαδή αργότερα με μια συγκεκριμένη πρόταση επί του θέματος. Ο λόγος για τον οποίο δεν την έχουμε διατυπώσει μέχρι στιγμή στην πρόταση αυτή, γιατί είναι πολύ πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Τα εθνικά συστήματα είναι πολύ πιο μεγάλης πολυπλοκότητας από το δικαίωμα αυτό καθ' αυτό πρόσβαση σε δικηγόρο. Αναφέρατε για παράδειγμα παρακαλώ πολύ εστέ σιωπηλή ενώ είστε μέσα στην αίθουσα. Κυρία Λεμπάιλ. Η κυρία Λεμπάιλ προσπαθεί να ολοκληρώσει την παρουσίασή της. Παρακαλώ πολύ. Ναι, λοιπόν, είναι φυσική άσκηση, γυμναστική για τις φωνητικές χορδές, λέει η κυρία Λεμπάιλ. Λοιπόν, για να επανέλθω στο ερώτημα, ήθελα να σας διευκρινίσω ότι μόνο στο 1 των περιπτώσεων ε, εποφελούνται τέτοια ε, αρρωγή. Πρέπει και αυτό να το έχουμε, αν θέλετε, σε οπτική, αλλά είναι ένα στοιχείο που, θα, που χρήζει περαιτέρω μελέτης, πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Θέσατε ερώτημα σε ό,τι αφορά την έρευνα στο χώρο κράτησης. Δεν ξέρω αν η λέξη έρευνα είναι σωστή. Ο δικηγόρος δηλαδή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες κράτησης δεν θα είναι τέτοιας φύσης ή υφής που θα θέτουν σε κίνδυνο τα θεμητά και νόμιμα δικαιώματα του πελάτη του. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε περισσότερα ερωτήματά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η συγκίτρια κυρία Αντωνέσκου ήθελε να κάνει κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις. Επιτρέψτε όμως να σας ζητήσω, να σας παρακαλέσω να το κάνετε σύντομα. για η ψηφοφορία που μεταφέρθηκε για τις 5 ε, και 4 Πολλοί από αυτούς θα ψηφίσουν ήδη παρόντες. Πρέπει να το έχουμε λοιπόν αυτό υπόψη μας. Και βέβαια, είμαστε ήδη καθυστερημένοι εδώ. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε υπομονή από την κυρία Λεμπάιλ, να γίνει η ψηφοφορία και μετά να συνεχίσουμε σε κοινή συζήτηση για το επόμενο σημείο της μέρης διάταξη. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνική θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε σήμερα. Θα ήθελα να πω μετά τη συζήτηση και τη δευτερολογία της κυρίας Λεμπάγη είναι προφανές ότι θα πρέπει να κάνουμε πολλές προσπάθειες για την έκθεση αυτή να μην βιαστούμε. Εγώ θα προσπαθήσω να καταθέσω πριν τα Χριστούγεννα το σχέδιο έκθεσής μου και θα είμαι πολύ ανοιχτή στις συστάσεις και προτάσεις των συναδέλφων, αλλά αυτό έχω στο μυαλό μου χρονοδιάγραμμα, να υποβάλω την έκθεση πριν τα Χριστούγεννα. Έχουμε καθυστερήσει, λέει ο Πρόεδρος. Θα έχουμε και δεύτερη συζήτηση αργότερα με την κυρία Λεμπάγ, Αλλά εκεί θα είμαι πολύ πιο αυστηρό στο χρόνο αγόρευση. Θα είναι πολύ πιο σύντομε οι παρεμβάσει. Γιατί σας άφησα ελεύθερους στην πρώτη συζήτηση και μερικοί μακρηγόρησαν. Αυτό δεν θα ισχύσει στη δεύτερη περίπτωση, στην κοινή συζήτηση του πακέτου για τα θύματα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα και παρακαλώ όσοι δικαιούνται να ψηφίσουν και όσοι είναι εδώ για να ψηφίσουν να, να μην απογοητευτούν και μετά θα έχουμε τη συζήτηση. Ψηφίζουμε μια στιγμούλα, μια στιγμούλα παρακαλώ. Τώρα αναγγέλλω την ψηφοφορία. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, του κυρίου Άλβαρο για, το ευρωπαϊκό, για την Ενίσα, την, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών. Η κυρία Χέντ, διαδικαστικό. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως δεν είμαι η μόνη που στερείται διερμηνία σήμερα συνεδρίαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε σουηδική διερμηνία. Είμαι και τακτικό μέλος της συνεδρίας. Έχουμε τόσο σημαντικά θέματα που μας απασχολούν σήμερα και είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε διερμηνία. Ξέρω ότι η αίθουσα είναι μικρή, δεν προβλέπει όλες οι καμπίνες, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η, Σουηδη... η βουλευτής ε, δεν ε, δικαιούται, δεν έχει διερμηνία. Λυπούμε πολύ γι' αυτό. Συγγνώμη, σας ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη και ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Πάντα το ίδιο συμβαίνει. Δυστυχώς η μόνη ελεύθερη αίθουσα για τη συνεδρίασή μας ήταν αυτή που προβλέπει μόνο 12 καμπίνες. Ήταν αδύνατο να εξασφαλίσουμε διερμηνία για όλες τις γλώσσες. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας, σημειώνουμε την παρατήρηση και περνάμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Άλβαρο Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Άλβαρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, Chair. Κύριε Πρόεδρε, μια και έχουμε πείσει χρόνο, δυστυχώς θα πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία λόγω του blackout. Δεν καταφέραμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και τώρα μας πιέζει ο χρόνος. Υπάρχουν επιφυλάξεις και στις, ε, στην τροπολογία 18 ο κατάλογος ψηφοφορίας έχει μείον για τις απαιτήσει ε, ως προς τον οργανισμό. Αυτό βλέπω σε, στις καταλόγους ψηφοφορίας δύο, ομάδων, δύο ομάδων. Παρακαλώ αναθεωρήστε γιατί μαζί με τον Κάρλος Κοέλιο για πρώτη φορά έχουμε ε, τον οργανισμό αυτό που θα συστηθεί ε, στο Τάλιν και το Στρασβούργο και βέβαια το Συμβούλιο θα καθορίσει την έδρα του οποιοδήποτε οργανισμού. Αυτό δεν αμφισβητείται, δεν είναι επίμαχο και το συζήτησε και το πρωί με τη Γραμματεία ε, και με τον εκπρόσωπο του, της Πολωνικής Προεδρίας ε, που κρίνει πολύ λογική την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σημείο αυτό. Και μια και είμαστε και συναρμόδιοι για τον προπολογισμό αρχή, θα πρέπει να δούμε το κατά πόσο τηρούνται οι προποθέσει για την έδρα. Υπάρχουν τέσσερα σημεία. Τοποθεσία, να είναι σε κεντρική τοποθεσία, να είναι ένα ενιαίο κτίριο που θα αφιερώνεται αποκλειστικά στη, στον οργανισμό αυτό και θα εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας δεδομένων. Και θα αποτελεί την πλέον αποτελεσματική απόψη κόστου λύση. Πολύ σημαντική προπόθεση εν μέσω χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Δεν λέμε πού θα α, τοποθετηθεί αυτή η έδρα. Και κανένα δεν θα πρέπει να έχει αφιβολίε για το ότι δεν είναι επιμάχο αυτό το θέμα. Όταν το δέχτηκε το Συμβούλιο την περασμένη φορά, εμεί καθορίσαμε κάποιε απαιτήσει που θα τοποθετηθει αυτη η εδρα και κανενα δεν θα πρεπει να εκπληρωθούν ε, μια αρνητική ψήφο σε, αυτό το σημείο θα ήταν ε, πολύ κακό μήνυμα προ το Συμβούλιο που δέχτηκε τη θέση του, του Κοινοβουλίου και ίσω επαναχωρήσει. Μια τέτοια επαναχώρηση θα αποδεσμεύσει και τη δική μα θέση στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει όταν συζητήσουμε άλλου οργανισμού και το τι περιμένουμε από αυτού. Θα ήθελα να υπενθυμίσω λοιπόν στους συναδέλφους ότι είχαν υπερψηφίσει αυτό το θέμα στον Οργανισμό Διαχείρισης ε, IT και, το, και πέρασε και στην Επιτροπή. Και μάλιστα θα τεθεί σε λειτουργία τόσο λίγο αυτός ο οργανισμός. Ε, είχαμε μερικές συναντήσεις με τους και με πολύ αγαστή συνεργασία και το βλέπω αυτό και στο κατάλογο της ψηφοφορίας. Γιατί νομίζω ότι όλοι μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο της έκθεσης. Ωραία, θα ψηφίσουμε. Ο κύριος Μπουσουτήλ σήκωσε το χέρι, θέλετε διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, αφεβάλλω αν το προηγούμενο σημείο ήταν διαδικαστικό. Ναι, αλλά είμαι εισηγητή, λέει ο κύριο ε, Αλβάρο. Ναι, αλλά ε, ο εισηγητή ε, έδωσε κάποιε συστάσει προ τι ομάδε. Μπορώ να απαντήσω πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. η έκκληση ο ο εισηγητή σε δύο πολιτικές ομάδες να αλλάξει το κατάλογο ψηφοφορίας τους. Ε, Σέβομαι πλήρω τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την επιλογή των εδρών των οργανισμών και το ΕΛΚ πιστεύει ότι οι προποθέσει ε, που θεσπίζονται στην τροπολογία Άλβαρο είναι πολύ ειδικέ και ουσιαστικά αποκλείουν τις ε, τις τωρινές τοποθεσίες αυτού του οργανισμού, τις τωρινές έδρες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αμφισβητείτε η επιλογή συγκεκριμένων ε, τοποθεσιών, συγκεκριμένων πόλεων για συγκεκριμένους οργανισμούς, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πραγματικά επικίνδυνο προηγούμενο. Γι' αυτό και έχουμε αρνητικό πρόσημο στο κατάλογο ψηφοφορίας. Κύριε Άλβαρο, θα ήθελα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ναι, δεν θέλω να κάνουμε διάλογο εδώ. Να υπενθυμίσω στο Σάιμον ότι η διατύπωση στην περίπτωση αυτή είναι ταυτόσιμη με παρόμοια έκθεση για τον οργανισμό επικοινωνίας και τεχνολογιών επικοινωνιών. Είναι ακριβώς η ίδια διατύπωση. Πού το πρόβλημα. Εντάξει, ψηφίζουμε συμβαστική τροπολογία ένα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Those again. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Ποιος είναι υπέρ. Ή μάλλον συμβαστική τροπολογία 2 λέει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, μου ξέφυγε λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική τροπολογία 2 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, τροπολογία 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. δεύτερο τμήμα της 37 γιατί είχαμε ψηφοφορία κατά τμήματα το πρώτο έχει καταπέσει δεύτερο τμήμα τώρα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές Μάλλον να εγκρίνεται. Δεν θέλει κανείς ηλεκτρονικό έλεγχο, εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 13, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτη παράγραφος που είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερη παράγραφος δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό Τροπολογία 44 έχει αποσυρθεί. Νόμιζα ότι 18 ότι μπορούμε να την ψηφίσουμε μια και δεν έχει ψηφιστεί 18. Λοιπόν, καλά, αποσύρθηκε. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογικέ σκέψει. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, αποσύρθηκε.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 την έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια ψήφος επιπλέον εκ μέρους του ΕΛΚ. Ποτέ δεν είναι αρκετές ψήφοι του ΕΛΚ, λέει ο κύριος Δεκάμπ. 48 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση του κυρίου Άλβαρο. Συγχαρητήρια κύριε Άλβαρο. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε την ψηφοφορία. Όσοι παραμείνουν στην αίθουσα παρακαλώ να μείνουν ήσυχοι και σιωπηροί και να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Λεμπάη για την υπομονή, την ιόβα υπομονή της. Τώρα περνάμε στην κοινή συζήτηση για δύο στοιχεία του πακέτου για τα θύματα. Παρακαλώ, επιμένω στο θέμα ησυχία.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 Ξανά, κύριε Λεμπάιλ, ευχαριστώ για την υπομονή σας και την κατανόηση της κατάστασης. Όπως συμβαίνει συνήθως με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, το πρόβλημα με το χρόνο, το να προσπαθούμε να προλάβουμε, είναι συνηθισμένο σας. Σας καλώ τώρα στην κοινή συζήτηση για αυτά τα δύο μέτρα, για τα θύματα, εσείς που σκοπεύετε να πάρετε το λόγο, να έχετε υπόψη όχι πάνω από δύο λεπτά. Δεν είχαμε χρονικό όριο για το πρώτο μέρος της συζήτησης και το ξεπεράσαμε. Κάναμε κακοδιαχείριση του χρόνου. Τώρα λοιπόν προσπαθούμε να προλάβουμε γρήγορα. Κυρία Λεμπάιλ, αρχίζετε την παρουσίαση, την κοινή παρουσίαση των ελάχιστων προτύπων για τα θύματα και για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και το σημείο 5, αμοιβαία αναγνώριση με τον προστασία σε αστικές υποθέσεις. Κυρία Λεμπάη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως είναι κατάλληλο τώρα αφού συζητήσαμε τα δικαιώματα των υπόπτων να συζητήσουμε στα δικαιώματα των θυμάτων. Καταλαβαίνετε ότι ε, αυτά συνδέονται. Όπως και η προσέγγιση που έχουμε. Τώρα, όσον αφορά τα θύματα. Αυτό που έχει προτείνει η Επιτροπή είναι δύο διαφορετικά στοιχεία στο ίδιο πακέτο. Το ένα είναι τα ελάχιστα πρότυπα για τα θύματα. Το άλλο είναι είναι το EPO. Έχει σχεδόν υιοθετηθεί και ευχαριστούμε πολύ το Κοινοβούλιο γι' αυτό. όσον αφορά τα ελάχιστα δικαιώματα για τα θύματα. Ποιο είναι το κίνητρο για αυτή την πρόταση. Τα θύματα πρέπει να τυχαίνουν μεταχείριση με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στην νομοθεσία και αυτή η νομοθεσία συνδέεται με την κατάρτιση που, είναι, που έχει πολύ μεγάλη σημασία σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζεται ένα θύμα στα κράτη-μέλη. Το πρώτο που κάναμε είναι να παρατείνουμε την έννοια του θύματος, να την επεκτείνουμε και να συμπεριλάβουμε και τα μέλη της οικογένειας σε αυτήν γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένα θύμα υποφέρει, υποφέρουν και τα μέλη της οικογένειας γύρω από το θύμα. γιατί θα ενδέχεται να χρειαστεί να πρέπει να φροντίσουν το θύμα, να τον βοηθήσουν και στη δικαστική διαδικασία και μπορεί να τύχουν και αυτό μπορεί να τύχει και αυτά να είναι αντικείμενο εκφοβισμού. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό να αφορά και τις οικογένειες, να έχουν και οι οικογένειες δικαιώματα ως θύματα. Οι οικογένειες τώρα των θυμάτων που έχουν επιζήσει. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη και προστασία. Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο στην ε, μεταχείριση των ε, θυμάτων που είναι προς όφελός τους. Η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη δεν είναι ίδια. Η σύστασή μας είναι να υπάρχουν, να πρέπει να υπάρχουν οργανισμοί υποστήριξη των θυμάτων σε κάθε κράτος μέλος ή αν δεν υπάρχουν να αναπτυχθούν. Όταν ερωτώνται τα θύματα, τις περισσότερες φορές απαντούν ότι δεν είναι σίγουροι για τα δικαιώματά τους, δεν είναι σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν και τι όχι. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι να, παρέχε, να παρέχονται πληροφορίες για τα δικαιώματά του στα θύματα και να διασφαλιστεί ότι αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται με τρόπο κατανοητό για το θύμα. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη μετάφραση και τη διερμηνία. Καθώς επίσης και να φροντίσουν τα πιο ευάλωτα θύματα, για παράδειγμα εκείνα που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Προτείνουμε επίσης, κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας, τα θύματα αυτά να έχουν απαραίτητη προστασία. Και πάλι εδώ συμπεριλαμβάνονται τα ευάλωτα θύματα, έτσι ώστε να μην υποφέρουν από περαιτέρω συναισθηματική φόρτιση. Υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν τα θύματα ιδιαίτερα ευάλωτα ή όχι. Ε, και εδώ αναφέρομαι στο γένος, στην ε, εθνότητα, στην, ε, στις σεξουαλικές προτιμήσεις. Φυσικά, τα θύματα ενδέχεται να είναι ευάλωτα ανάλογα με τα δεινά που έχουν υποστεί, για παράδειγμα με οικογενειακή βία ή τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θέλουμε να συμπεριλάβουμε και γι' αυτό ζητάμε από τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν το βαθμό κατά τον οποίο στον οποίο είναι βάλωτα τα θύματα από τον είναι βάλωτα στον εκφοβισμό, στον εκφοβισμό κατ' επανάληψη, όπως για παράδειγμα στην οικογενειακή βία. Ή τον εκφοβισμό κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας. Αυτό που επίσης συνειδητοποίησαμε είναι ότι αυτό θα πάρει χρόνο και ότι στη διάρκεια της ε, διαδικασίας αυτής το θύμα πρέπει να είναι προστατευμένο. Αυτή όμως η προστασία, εάν για παράδειγμα το θύμα αποφασίσει να πάει σε κάποιο άλλο, άλλο κράτος μέλος, μπορεί να χαθεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε την ε, εντολή προστασίας στις αστικές υποθέσεις, η οποία είναι συμπληρωματική του κανονισμού του ΥΠΙΟ για τις ποινικέ υποθέσεις. Αυτό προτείνουμε, με λίγα λόγια. Κάτι θα ήθελα να προσθέσω. Η οδηγία επίσης διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν ε, μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και θα υπόκεινται στην απόφαση των δικαστών. Τα μέτρα αυτά θα προστατεύουν τα δικαιώματα των θυμάτων και των υπόπτων. Στην ουσία αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι όλες οι πλευρές θα απολαμβάνουν σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεμπάιλ. Ευχαριστώ που ήσασταν σύντομοι και περιεκτικοί. Τώρα αρχίζουμε τη συζήτηση. Την αρχή θα κάνουν οι δύο εισηγητές. Σερίλ και Ρομέρο. Και μετά η συζήτηση θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής. Δύο λεπτά. Η κυρία Χιμένες Δεσερίλη, πρώτη μας συγγήτρια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι θα είμαι λακωνική, μια και παρατάθηκε η προηγούμενη συζήτηση και πήρε κάποιο το χρόνο της δικής μας. 75 εκατομμύρια θύματα βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα άξιζαν λίγο περισσότερο χρόνο συζήτησης. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μπάιχ γιατί ξεκίνησε την ομιλία της με τον όρο αξιοπρέπεια. Θα ήθελα επίσης να πω ότι με τη χρήση του όρου αυτού της αξιοπρέπειας κατάλαβε τον κόσμο των θυμάτων και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτή την πετυχημένη οδηγία που προβλέπει κάποια ελάχιστα πρότυπα για δικαιώματα, υποστήριξη και προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Και θα ήθελα να επιδοκιμάσω και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή την οδηγία, γιατί μια τέτοια οδηγία χρειαζόμασταν κατεπηγόντω στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα βοηθήσει όχι μόνο τα θύματα πάση μορφή βία, αλλά θα διατρανώσει την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόκειται για μια οδηγία που θα βελτιώσει την εικόνα και την ιδέα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αυτή ε, βλέπει το φως μετά από την έγκριση που έγινε πριν από μία εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας, που μετά από πολλές δυσκολίες ε, ευωδόθηκε μαζί ε, με τα δύο εντάλματα για αστικέ και ποινικέ υποθέσει. Έτσι θα βοηθήσουν περισσότερα τα θύματα. Για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσεγγίσει με οριζόντιο τρόπο αυτό το φαινόμενο, προκειμένου να εξασφαλίσει τα θύματα αυτά μία μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ενισχύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα διάφορα δικαιϊκά συστήματα και διευκολύνεται η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που είναι ως λίθος του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Καθορίζονται στην οδηγία αυτή διάφορες κατηγορίες θυμάτων ανάλογα με το είδος εγκληματικής πράξης που υπέστησαν ή από τις ειδικέ προστα... Ε, περιστάσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Η ανακοίνωση που χρησουν ιδιαιτερης προστασιας Επιτροπής κάνει ειδική μνήμα των θυμάτων τροχαίων, των θυμάτων της τρομοκρατίας, των ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων, δηλαδή ανήλικα άτομα, ανάπηροι και θύματα σεξουαλικής βίας ή θύματα σωματεμπορίας. Επίσης προσδιορίζονται πέντε επίπεδα προστασίας με αντίστοιχα νομοθετικά όργανα. Αναγνώριση και ε, αξιοπρεπής μεταχείριση, αποκατάσταση ε, αποζημίωση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κατεπηγόντως αυτήν την οδηγία γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμη προκειμένου να βοηθήσουμε τα θύματα της βίας. Και μάλιστα δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο όραμα για τη σημερινή κατάσταση, ούτε μια συγκεκριμένη εντύπωση. Όταν μιλούμε για την βία μεταξύ των φύλων, δεν έχουμε καν στατιστικά στοιχεία, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερε στατιστικέ πληροφορίε και βάζει δεδομένο για να ξέρει τι μέτρα χρειάζονται και πώς αναδράσει. Θα ήθελα τελικά να υποβάλω και μερικές ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το περιεχόμενο τη Οδηγία. Το θέμα του ευάλωτου χαρακτήρα των θυμάτων αποτελεί σημείο κλειδί της ε, οδηγίας. Αναφέρθηκαν τα θύματα σεξουαλικής βίας και τα θύματα ε, σωματεμπορίας, ε, τα ανήλικα άτομα, τα ανάπηρα άτομα, ως ιδιαίτερα ευάλωτα. Υπάρχουν όμως και θύματα άλλων εγκληματικών πράξεων και άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών. Δεν θεωρείτε ότι και άλλα θύματα μπορεί να είναι ευάλωτα. Γιατί επιλέξατε ορισμένε μόνο κατηγορίες ευάλωτων ατόμων. Δεύτερη ερώτηση. Η ανακοίνωση που λάβαμε μαζί με την οδηγία αναφέρει ως πρώτο είδος ευάλωτων θυμάτων τα θύματα της τρομοκρατίας. Στην αιτιολογική σκέψη, στο άρθρο 18 γίνεται λόγο των θυμάτων τρομοκρατία. Αντίθετα, η οδηγία στο άρθρο 18 δεν αναφέρει τίποτα για τα θύματα της τρομοκρατίας. Παραλείπονται τελείω από το άρθρο της οδηγίας. Γιατί? Στην οδηγία πλαίσιο που αφορά το καθεστώς του θύματος στην δικονομική διαδικασία του 2001 περιλαμβάνεται ο ορισμός της έννοιας του θύματος. Πολλές διατάξεις αποφάσεων αναφέρονται στην περίπτωση του ευάλωτου θύματος. Γιατί η συγκεκριμένη οδηγία δεν μας δίνει τον ορισμό του ευάλωτου θύματος. Είναι πολύ σημαντικό τα δικαιώματα και η υποστήριξη στα θύματα να στηρίζονται στις ατομικές ανάγκες του κάθε θύματος. Για παράδειγμα, κάθε θύμα έχει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με το τι έγκλημα υπέστη και τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διανύουμε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι ζωτική σημασία κάθε κράτος μέλος να εντοπίζει σε ποιε καταστάσεις χρειάζονται περισσότεροι πόροι και εκεί να τους αφιερώνει. Είχαμε πολλά προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία. Φαντάζομαι και αυτή η οδηγία ίσω προσκρούσει σε προβλήματα στο Συμβούλιο. Ίσως τα κράτη-μέλη δείξουν επιφυλάξει ή μήπω τελικά θα καταλάβει το Συμβούλιο ότι η ικανοποίηση του θύματος θα αποτελέσει κέριο παράγοντα για την ανάρρωση, για την ανάνυψή του, την αποκατάστασή του και θα είναι κάτι που θα μας οδηγήσει και σε οικονομία σε τελική ανάλυση. Για μένα είναι μεγάλη μέρα σήμερα, γιατί από τότε που ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσα ότι υπήρχαν πολλά κενά στο δρόμο μας να βοηθήσουμε τα θύματα και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για την έκθεση αυτή. Κύριε Ρομέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Λεμπάη για τις εξηγήσει που μας έδωσε παρόλο που είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτά τα δύο θέματα για αυτή την οδηγία δηλαδή και τον κανονισμό που αφορά το, την Ευρωπαϊκή Εντολή προστασίας για αστικέ υποθέσεις. Βέβαια, κατ' ουσία αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Πάντως, ο κανονισμός έχει το πλεονέκτημα ότι είναι άμεση εφαρμογή και θα εφαρμοστεί πολύ γρήγορα στις χώρες που ε, ε, είναι δυνατή μια τέτοια εφαρμογή. Οπότε η πρώτη ερώτησή μου είναι η εξής. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει ήδη, έχετε συντάξει ένα των χωρών που επηρεάζονται από τον κανονισμό, γιατί πρόκειται για αστικά μέτρα, μέτρα αστικού δικαίου. Οπότε όταν ε, ε, η δικαιοδοσία δεν είναι δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων ποινικών, τότε εφαρμόζεται η οδηγία. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η οδηγία που αναφέρεται στις ποινικέ υποθέσεις θα εφαρμοστεί πολύ αργότερα. Γιατί θα πρέπει πρώτα να ενσωματωθεί στι εθνικέ νομοθεσίε. Δεν είναι άμεση εφαρμογή όπω ο κανονισμό. Χαιρόμαστε για την επιτάχυση των διαδικασιών αυτή τη οδηγία και δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη συζήτηση στον κανονισμό. Έτσι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να μεταφέρουν την οδηγία αυτή στις εθνικές νομοθεσίες πολύ πιο γρήγορα. Και κατά τη γνώμη μου αυτή η διαδικασία θα είναι μια διαδικασία αξιολόγησης. Είναι φυσικά λογικό να επικροτούμε αυτόν τον κανονισμό και στη διάρκεια της συζήτησης θα αναλύσουμε πιο λεπτομεριακά τη θέση μας για τα επιμέρους ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρομέρο. Τώρα άρχεται η συζήτηση. Σας υπενθυμίζω ότι το δίλεπτο είναι κανόνας απαράβατος, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Κυρία Μπάουερ πρώτα. Köszönöm szépen, elnök úr. Én két kérdést szeretnék föltenni az előterjesztőnek. Az 5. és a 15. cikkei fordítás. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το κόστος μετάφρασης θα το αναλαμβάνει ποιο, ποια πλευρά. Είμαι στα δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε. Υποθέτοντας λοιπόν ότι υπάρχει μια εξομάλυνση το κόστος, γιατί θα πρέπει να γίνει μετάφραση όταν την όλη, σε σχέση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τώρα, απόφαση στο σημείο 16 τον εποφελείται από το πλέον, ε, όπως αναφέρει, εποφελούμενο από το πιο εποφελές ε, νομικό καθεστώς. Όλο αυτό το παράθεμα. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε μεγαλύτερη ε, ακρίβεια για κάλυψη του σημείου αυτού. Γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση του θύματος μπορεί να είναι πολύ διαφορετική σε συνάρτηση με τη χώρα στην οποία βρίσκεται. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο άρθρο 16. Θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι και να κάνω μια ερώτηση. Μιλάμε για το δικαίωμα των θυμάτων και φυσικά και αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα όμω και εγώ να υπενθυμίσω για την ποινική διαδικασία. Η ποινική διαδικασία είναι μια διαδικασία όπου συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, εάν έχει διαπραχθεί ένα ποινικό αδίκημα. Δεύτερον, ποιος είναι ο δράστης και ποιο είναι το θύμα. Έχουμε δύο ορισμούς του δράστη. Ο κατηγορούμενος και ίσως ο δράστης. Για το θύμα υπάρχει μόνο ένας ορισμός και αυτό κάνει τη συζήτηση δύσκολη. Πιστεύω ότι για τα θύματα είναι σημαντικό να, υπάρχει, ε, ε, να έχουν ενεργό ρόλο στην ποινική διαδικασία, να πληροφορούνται για το τι συμβαίνει, για, την, ε, για το καθεστώς της ποινικής διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν και εκείνα να δουν τι επιπλέον βήματα μπορούν να κάνουν ως θύματα. Επίσης με αυτή την οδηγία πιστεύω ότι όπου υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Πολλά θύματα όταν ο δράστης πραγματικά καταδικάζεται δεν έχουν πλέον καμία βοήθεια όταν προχωρούν σε αστικές, σε, δικ, αστικού περιεχομένου. Τι γίνεται λοιπόν στην ε, οδηγία με αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε συμμερίζομαι αυτό που είπε στην αρχή η Αφιερώσαμε σχεδόν μια μισή ώρα στην προηγούμενη συζήτηση. Με κάθε σεβασμό όμως δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που γίνεται λόγος για την προστασία των θυμάτων να το πραγματευόμεθα σαν ένα θέμα, αν θέλετε, συμπληρωματικό, επικουρικό ή επιφανειακό είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε κάθε φορά να δίνουμε μια μισή ώρα για την προηγούμενη συζήτηση για κάθε κάτι άλλο. Θα πρέπει κάθε φορά να κάνουμε πριν συζήτηση του πώ θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Η κυρία Λεμπάιλ είπε ότι είναι μια συνάντηση για ύστερη φάση λόγω ψηφοφορία. Μα έδωσε, είχε την ευγένεια να μα δώσει επιπρόσθετο χρόνο. Ναι, μα η προηγούμενη συζήτηση και οι δύο μαζί αυτή τη στιγμή. πρόεδρο και βουλευτής Παρακαλώ πολύ κύριε Αλθάνο. Δεν είναι δυνατόν να... να θέμα. Τα θέματα προστασίας των δικαιωμάτων, προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, όπω και όλων των δικαστικών, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δεν σα καταλαβαίνω. Παρακαλώ που να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο για να κάνετε την παρέμβασή σα. Όχι με το δικαστικό. Όχι, δεν ήταν μια, ε, ένα παράπονο, είναι διαπίστωση. Γιατί οι προηγούμενοι μιλούσαν πριν από 10 λεπτά, χωρί να είναι εισηγητέ. Ήθελα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πω στην κυρία Λεμπέιθ, στην ε, έκθεσή μου σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο παρουσιάστηκε, υποβλήθηκε και υπερψηφίστηκε ομοφόνο στην Επιτροπή Ελευθερίων την περσμένη εβδομάδα, ζητήσαμε κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα είχε στόχο η να υπάρχει προστασία μαρτύρων και των ε, οικογενειών του σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Και για κάθε τυπολογία ε, θυμάτων, είτε θυμάτων από οργανωμένη εγκληματικότητα, τρομοκρατίε ε, ή οτιδήποτε άλλου είδου. Χρειάζεται λοιπόν η προστασία των μαρτύρων από τη δικαιοσύνη. Και αυτό ξεπερνά την όλη διαδικασία των δικαστικών δια... διαμάχης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια ενδεχόμενη επέκταση της οδηγίας που συζητάμε σήμερα. Κύριε Κίκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο Προφανώς ε, πλέον τα πράγματα ε, σκληραίνουν. Θα ήθελα καταρχάς να πω και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όντω χρειαζόμαστε πολύ υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων. Είμαι σχετικά ευτυχή για το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχετικά καλό ιστορικό στο θέμα αυτό. Όμω, και το τονίζω αυτό το όμω, είναι σαφέ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Δεν θέλω να δω εναρμόνιση των δικαιωμάτων, αλλά θέλω να δω κάποιο αντίστοιχο ε, προστασία των θυμάτων. Και αυτό μπορεί να μα φέρει σε αυτό το σημείο. Δεν είναι νομίζω δυνατόν να παραβλέψουμε τα εθνικά δικαιϊκά συστήματα, εθνικά ποινικά συστήματα όπου υπάρχει κάποια σχετική προστασία, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον ως Επιτροπή και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουμε προσεκτικά την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το οικονομικά προσιτό των προτάσεων αυτών, νομίζω θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι τροπολογίες τις οποίες συζητάμε εδώ να είναι προσιτέ για να μην χάσουμε το όλο θέμα απλά και μόνο για λόγου οικονομικού κόστου. Και ένα τελικό σημείο. Η οδηγία αυτή, κύριε Πρόεδρε, θα καλύψει μόνο τον Ευρωπαίο πολίτη σε χώρα μέλος ή σε ευρύτερο έδρος και έναν Βρετανό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αντιστρόφω ένα Αμερικανό στο έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωση θα καλύπτεται από αυτή την νομοθεσία. Πρέπει να είμαστε σαφείς πάνω σε αυτό και γενικά σα υποστηρίζω επί του θέματος. Ευχαριστούμε. Κύριος, ε, ε Αγγελίλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί προφανώς υπάρχει απειροελάχιστος χρόνος να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Θα ήθελα να πραγματευτώ ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που ε, ήταν ιδιαίτερα προσφυλές και στην Επίτροπο Ρέντινγκ. Το να αφιερωθεί, δηλαδή να δοθεί ιδιαίτερη, ιδιαίτερη ε, προσοχή στους ανηλίκους. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της όλης ποινική διαδικασίας, να δοθούν ε, εγγύησης πλήρη ευρέως φάσματος σε ό,τι αφορά την προστασία του προσώπου, του τρόπους και τις διαδικασίες ανάκρισης και σε ό,τι αφορά το, τη διάρκεια των διαδικασιών, γιατί οι ανήλικοι είναι πρωτίστως τα πλέον ευάλωτα θύματα και που κινδυνεύουν διπλή θυματοποίησή τους και την αρχική του ότι είναι θύματα κάποιου εγκλήματος και δευτερογενώς γιατί είναι θύματα ενός ποινικού συστήματος, ενός συστήματος ε, ποινικών διαδικασιών που μπορεί στη συνέχεια να παρεμβαίνει αρνητικά στην ψυχολογία και στην προσωπικότητα του ανηλίκου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά. Κύριε Σκοτσέτα. Ναι, ευχαριστώ όντω να τα καταφέρω σε δύο λεπτά. Ίσως και να, έχω και λίγο περισσότερο, να χρειαστώ λίγο περισσότερο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Αλφάνο όταν έθεσε το πλέον γενικό ευρύ θέμα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα αυτών που προσάγονται στη δικαιοσύνη αυτών των μαρτύρων σε περίπτωση τρομοκρατίας. Δύο σκέψεις όμως που θεωρώ πολύ σημαντικέ. Ορισμένε φορέ πεθαίνουν, σκοτώνονται θύματα δηλαδή δεν είναι θύματα μόνο στη διάρκεια διαδικασιών. Πολύ συχνά τα θύματα πλέον είναι οι οικοί του θύματος. είναι τα παιδιά, η σύζυγος, σκεφτείτε όλους αυτούς τους δικαστικούς που έχουν δολοφονηθεί, τους αστυνομικούς που έχουν δολοφονηθεί στις τρομοκρατικές επιθέσεις ή επιθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Και στην πολιτική έχει υπάρξει ε, δολοφονία στη μάχη αυτή, αν θέλετε, καταπώνησης και κατάτος του ηθικού. Μας οδηγεί λοιπόν αυτό το θέμα στο ζήτημα του τι πρέπει να κάνουμε σχετικά. Σας λέω σχηματικά, αφενός έχουμε το θύμα, το άτομο, και από την άλλη τον επιτιθέμενο ως ε, θύμα επίσης. Ορισμένες φορές διευρύνεται το μοντέλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να βρούμε στο σχήμα αυτό την εξωτερική απειλή, την απειλή της τρομοκρατίας, γιατί πολύ συχνά στο μοντέλο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν συνδέονται οι μετασχηματισμοί οι οποίοι έχουν επέλθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δει σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα με την παγκοσμιοποίηση αυτού του φαινομένου και πώς το φαινόμενο αυτό ε, ιδιαίτερα ανησυχητικό σε κάποιες χώρες. Σε κάποιες χώρες όπως στην πόλη μου για παράδειγμα, το πρόβλημα είναι από το 87 μέχρι το 90 δολοφονήθηκαν 300 άτομα σε αυτή την, στον πόλεμο, τον ακήρυκτο πόλεμο της μαφίας. Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε στην Ελβετία, την Αγγλία, τη Γαλλία, θα είχε τύχει της προσοχής ποιος ξέρει πόσο διεθνών οργανισμών έχουν δολοφονηθεί, για παράδειγμα, όπω μια νοικοκυρά που κάποια μέρα πήγε για ψώνια, πήγε στο σούπερ μάρκετ και απλώ βρέθηκε να αγοράζει, να αγοράζει φρούτα από κάποιον ο οποίο υπήρξε θύμα ε, επίθεση μαφιόζου και την πήραν και αυτή τα σκάλια. από τις χώρες, σε κάποιες από τις χώρες υπάρχουν τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα όμως του οργανωμένου κλιματικότητας είναι πραγματικό και αυτό. Το πρόβλημα των ε, μαρτυρίας υπόπτων στην δικαιοσύνη είναι πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα για να υπάρξει οικονομική υποστήριξη στα οικογένειε των θυμάτων. Ποιες είναι οι εγγύσεις. Εκτέω ε, θα ήταν να έχουμε σχετική συνεννόηση και με τη ΣΥΠΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να φτάσουμε σε μια συνθήκη καταρχάς μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι την προστασία που δίνεται σε κάτι που σκοτώσει 100 άτομα. Πρέπει να αλλάξει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Υπόθηκαν πολλά σωστά πράγματα. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Θα ήθελα δύο ερωτήματα να θέσω. Πρώτον, όσον αφορά τους ορισμούς, τον ορισμό του θύματος, που έχετε ήδη μια ευρύτερη προσέγγιση που συμπεριλαμβάνετε τα μέλη της οικογένειας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα ήταν δυνατόν ή λογικό να παρέχετε νομική αντιπροσώπευση. Θα ήταν δυνατό, δυνατόν να συμπεριληφθεί και αυτό στον ορισμό. Επίσης, όσον αφορά τις οντότητες που θα δρούν εκ μέρου των θύματων στι ποινικέ διαδικασίε. Αυτό δηλαδή το κείμενο, αυτό θα θέλαμε να πούμε. Το, η δεύτερη ερώτηση είναι για το νομικό καθεστώ των θυμάτων. Εμεί ω πράσινοι πιστεύουμε ότι το νομικό καθεστώ ε, λογικά δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο όσον αφορά τα συμφέροντα των θυμάτων. Επομένως, θα ήταν λογικό να ελαχιστοποιήσουμε ίσως τις συνθήκες ε, κάτω από τις οποίες θα μπορούσαν να υποφεληθούν τα θύματα. Για παράδειγμα η άδεια παραμονής που είναι περίπου ένας χρόνος. Αυτό θα ήταν λογικό πιστεύω. Τέλος. Ειδικά στο θέμα της διάκρισης, των διακρίσεων. Η βία, για παράδειγμα, που προκύπτει από ρατσιστικά κίνητρα. Είναι δυνατόν για οντότητες ή για νομικούς αντιπροσώπους να αντιπροσωπεύουν τα θύματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φως. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την πρόταση. Είναι περιεκτική για όλη την Ευρώπη και δίνει στα θύματα μία φωνή. Ήδη κάνατε λόγο για, τους, ε, για τις ενώσεις των θυμάτων. Στα εκτιμώντας όμως, στο εκτιμώντας 25, όσον αφορά την εθελοντική και όχι μόνο την επαγγελματική βοήθεια. Επίσης, όπως είπε η κυρία Ζίπελ και ο Τίμωθη, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των θυμάτων στις δικαστικές, ε, στις δίκες, είναι, θα πρέπει να βρίσκονται τα θύματα εκεί. πρέπει να προσέξουμε να μην διαταραχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην υπεράσπιση και στην ε, δίκη και στον, και κατηγορούμενο. Η έννοια του θύματος θα μπορούσε επίσης Έπειτα, στο άρθρο 12 θα μπορούσε να, να προσθεθεί το κόστος. Έπειτα στο άρθρο 18 την ανάγκη προστασίας του θύματος που πρέπει να αξιολογηθεί. Τι σημαίνει αξιολόγηση. θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτό το σημείο. Και το άρθρο 23. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο την διατύπωση και να πούμε από τύπος γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης. Κυρία Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπά για την παρουσίαση. Θα είμαι λακωνική γιατί με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους ότι το κείμενο είναι πολύ σημαντικό και η, ερμηνεία του, η διασταλτική ερμηνεία του ορισμού του θύματος είναι κάτι σημαντικό. Θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περαιτέρω, πάντως η αρχή είναι πολύ καλή. Αναφέρονται οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για το ότι δεν καταλήξαμε, δεν συμφωνία μετά από τη μακροχρόνια συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και, και τη διάκριση μεταξύ αστικών και ποινικών υποθέσεων. Ξέρω ότι το θέμα είναι και πολύ σύνθετο και περίπλοκο και ευαίσθητο, αλλά ενδιαφέρον θα ήταν να υπήρχε συμφωνία. Και μάλιστα και εσείς στην παρουσίασή σας, κύριε Λεμπάγη, μιλήσατε για την παράταση της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας μεταξύ της χώρας έκδοσης και της χώρας εκτέλεσης. Ε, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι ευκταίο και υπό το πρίσμα των θυμάτων. Ναι και μας πιέζει ο χρόνος, δύο σύντομες παρατηρήσεις. Ένα θέμα που αφορά τη σταθερότητα του νομικού καθεστώτος και το θέμα της αφήνειας ή της ε, ευκολίας πρόσβασης του κειμένου. Και πώς θα γίνει ο σχετισμός μεταξύ των εφιστάμενων μέσων και του νέου κειμένου για την προστασία των θυμάτων. Πώς θα γίνει ο συνδυασμός μεταξύ τους. Το κείμενο αυτό θα είναι μια οριζόντια οδηγία, σε αυτό προσβλέπει τουλάχιστον. Οπότε εστερνίζομαι και εγώ τις Ερωτήσει και επιφύλαξη των συναδέλφων. Φυσικά κάτι τέτοιο θα δώσει μεγαλύτερη προβολή και θα διευκολύνει την πρόσβαση στα δικαιώματα αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε στα, στην πρόταση και τα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και τα θύματα της τρομοκρατίας. Γιατί είμαστε οι περισσότεροι υπέρ της συμπερίληψης και των θυμάτων της τρομοκρατίας στην πρόταση αυτή. Κυρία Λεπάιλ, όσο και η συγκήτρια μας υπενθύμησαν ότι την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε ομόφωνα σε αυτή την Επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων υπέρ της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Εντάλματος Προστασίας που να επιτρέπει στα άτομα που είναι θύματα σε ποινικέ διαδικασίες να επωφελούνται προστασίας πέρα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το ένταλμα. Αυτή η ομόφωνη ψήφος αντικατοπτρίζει κατά την άποψή μου το πόσο σημαντική είναι η προστασία των θυμάτων για την Επιτροπή μας. Γι' αυτό και θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας μου να καλωσορίσω την παρούσα πρόταση της Επιτροπής η οποία υιοθετεί μια ευρεία προσέγγιση ως προς τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα τους περιεκτικούς ορισμούς όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας, τους συντρόφους και τα ευάλωτα θύματα. Προσβλέπουμε μια καλή συνεργασία με την εισηγήτρια, η οποία έχει μια πολύ δυνατή προσωπική και επαγγελματική δέσμευση ως προς τα θύματα εγκληματικών πράξεων, ώστε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση και την ενίσχυση του ευρέως χαρακτήρα της οδηγίας. Για εμάς είναι επίσης σημαντικό να εισαγάγουμε ορισμένες διατάξεις που να περιγράφουν συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης που θα πρέπει να παρέχουν τα κράτη-μέλη στα θύματα, όπως για παράδειγμα τα καταφύγια.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 ακόμα και αν το κράτος ζητήσει ε, να επανόρθωσει. Το κράτος δηλαδή πρέπει να καταβάλει αποζημίωση και να επανορθώσει τη ζημιά. Στο για παράδειγμα στην Ουγγαρία η σοσιαλιστική κυβέρνηση διέπραξε ε, όταν υπήρξε κάποιο έγκλημα το, δικαι... το κράτος έπρεπε να ε, προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωση εφόσον το κράτος δεν προχώρησε σε διαλεύκανση των εγκλημάτων τα οποία ε, είχαν συγκεκριμένα θύματα. Δυστυχώ στην Ουγγαρία είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα αυτά, είναι καθημερινά, διότι το κράτος είναι ασυνεπές ή αν θέλετε κατά συνεπή τρόπο δεν προχωρά στην διαλεύκανση εγκλημάτων. Θα είμαι πολύ σύντομη κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν είμαι θετική επέναντι στην πρόταση αυτή. Στις κάτω χώρες πριν από κάποια χρόνια το κόμμα μου εισήγαγε κάποιο παρεμφερή νομοθεσία. Θα ήθελα όμως να κάνω μια παρατήρηση περισσότερο φιλοσοφικής υφής, απειχώντας λίγο αυτά που είπε και η κυρία Σίπουλος προηγουμένως. Ε, ε, στο, τέλος, ουσιαστικά, ο καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης των θυμάτων είναι να υπάρχει ένα σωστά λειτουργών δικαιικό σύστημα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε την κακή λειτουργία της ε, δικαστικής εξουσίας στα κράτη-μέλη, παρέχοντας υπερβολικά δικαιώματα στα θύματα. Θα πρέπει να προστατεύονται από τα θύματα, από το ε, δικαιικό σύστημα και θα πρέπει όντως να απονέμεται δικαιοσύνη. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε να συζητάμε για περαιτέρω δικαιώματα. Ευχαριστούμε κυρία Έντβελτ. Τώρα λόγω και πάλι κυρία Λεμπάη και την ευχαριστούμε θερμά γιατί μας παραχώρησε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Αλλά πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λεμπάκη, δεν ξέρω αν θέλει εκπρόσωπο τη Πολωνική Προεδρία να κάνει ένα σύντομο σχολιασμό. Και τον θέλω να παρακαλώ να είναι λακωνικός ή λακωνική. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστούμε για το δίλεπτο που μου παραχωρείτε παρά το φορτωμένο σας πρόγραμμα. Η προστασία των θυμάτων αποτελεί προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας, προτεραιότητα που ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία που επετεύχθη στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης. Μέχρι στιγμής ε, το έργο του Συμβουλίου επικεντρώθηκε στην πρόταση οδηγίες για, το για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας σε ποινικέ υποθέσεις. Χάρη στις κοινέ προσπάθειες του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία, σε πολιτική συμβαστική λύση για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Και η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η αγαστή εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια του τριμενούς διαλόγου αποτέλεσαν σημαντική συνεισφορά και βοήθησαν ανεκτήμητα την Πολωνική Προεδρία να επιτελέσει αυτό το δύσκολο έργο της επίτευξη συμφωνία. Η οδηγία που θεσπίζει κάποια ελάχιστη ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα, υποστήριξη και προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων είναι σημαντική. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική εξέταση αυτής της πρότασης. Ως εκ τούτου, η Πολωνική Προεδρία θα υποβάλει εντός ολίγου αναθεωρημένη πρόταση για περαιτέρω συζήτηση και εξέταση στο Συμβούλιο. Ευελπιστούμε ότι θα εξετάσουμε ορισμένα ζητήματα αυτού του πακέτου στο επόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών τον Οκτώβριο. Και πιστεύω ότι από τη ζήτηση αυτή θα προκύψουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και θα καθοδηγήσουν το μελλοντικό έργο του Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διάφορες επιφυλάξεις και να συμφωνήσουμε σε μια γενική προσέγγιση. Προσβλέπω στη συνέχιση της καρποφόρας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πακέτο αυτό και σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε το Συμβούλιο. Κύριο Σελήνο, ζητώ συγγνώμη. Λυπάμαι, είχατε ζητήσει και εσείς το, είχατε ζητήσει και εσείς το λόγο, συγγνώμη. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα ελέγξαν από τους συναδέλφους που προηγήθηκαν. Ήθελα μόνο να κάνω μια παρατήρηση. Ε, κατ' εμέ τονίσαμε ιδιαίτερα τον ορισμό του, του εγκλήματος παρά του θύματος. Θα ήθελα να δώσουμε πολύ περισσότερο προσοχή στην κατάσταση και στον ορισμό του θύματος. Γιατί αν θέλετε ουσιαστικά περιγράφοντας τα εγκλήματα μπορούμε πάντα να αφήσουμε κάποιον απ' έξω είναι κάπως ενδεικτικός ο έλεγχος, αν θέλετε. Οι μαρτυρίες της ε, δικαιοσύνης αναφέρθηκε από κάποιους. Το, ο μάρτυρας δικαιοσύνης δεν είναι, αν θέλετε, ε, θύμα κάποιου εγκλήματος, αλλά είναι θύμα, αν θέλετε, του ίδιου του φουθάρους του, αν θέλετε, και της παρησίας του να βρεθεί. Επομένως, σας αφήσουμε απ' έξω τους ε, μάρτυρες ε, στη δικαιοσύνη, οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη. Θα πρέπει να εξατομικεύσουμε πολύ περισσότερο τον ορισμό του θύματος παρά εκείνον του ορισμού του εγκλήματος. Κυρία Λεμπάγη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πληθώρα ερωτημάτων που τέθηκε μετά από αυτή την πολύ συναρπαστική συζήτηση. Να σα ευχαριστήσω καταρχήν θερμά για την υποστήριξή σα, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι η πρόταση είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει πραγματικά να αφιερώσουμε την προσοχή μα στα θύματα, το ίδιο αν όχι περισσότερο από ό,τι στου υπόπτου. Και παρόλο που θα έχουμε ευκαιρία να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ε, χαίρομαι για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η βάση, το θεμέλιο για όλα αυτά είναι εύρυθμα δικαιικά συστήματα και σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Ακόμη όμως και μία εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να ξεχνά τα θύματα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προστασία, όπως και να έχει το πράγμα, στα θύματα. Πολλές ερωτήσεις ε, περιστράφηκαν γύρω από το κόστος και ποιος θα αναλάβει αυτό το κόστος. Θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα για το πιθανό όφελος μια σωστής μεταχείρισης των θυμάτων. Γιατί είδαμε τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Δυστυχώς ε, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό της ε, ενδοοικογενειακής βίας που κοστίζει στα κράτη-μέλη μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και η μελέτη υπολόγισε ότι η συνδρομή στα θύματα που δίνεται από την κοινωνία θα ήταν λιγότερο από 100, οικονομίες πάνω από 100 εκατομμύρια σε σχέση με το συνολικό κόστος. Βέβαια, 100 εκατομμύρια σε σχέση με τα 10-20 δισεκατομμύρια δεν είναι και πολλά. Αλλά είναι παρόλα αυτά μια συμβολή στη μείωση του γενικού κόστους της βίας. Βέβαια, θα χρειαστούν κάποια χρήματα για να δοθεί αυτή η ιδιαίτερη προσοχή προς τα θύματα. Αλλά αν τύχουν σωστή μεταχείριση στα θύματα, το συνολικό κόστος θα μειωθεί στο μέλλον. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν και για το οργανωμένο έγκλημα. Κατά την ε, σύνταξη της πρότασης, υιοθετήσαμε μια οριζόντια προσέγγιση για τα θύματα – όλα τα θύματα λαμβάνονται υπόψη και κατά τη γνώμη μου τα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος καλύπτονται από την πρόταση. Βέβαια, αν εσείς θεωρείτε ότι δεν αναφέρεται αυτό ρητά, ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ και την ανακοίνωση και το νομικό κείμενο και αν δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι καλύπτονται και τα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος, τότε θα μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Αναφέρθηκε μια ερώτηση για την προστασία των παιδιών. Αν ρίξετε μια ματιά στο άρθρο 18, διαπιστώνετε ότι υπάρχει ειδική μνήα των παιδιών. Τα παιδιά αναφέρονται ρητά ως ευάλωτα θύματα. Και φυσικά θέλουμε να τύχουν σωστής φροντίδας και μεταχείρισης τέτοια ευάλωτα θύματα όπως είναι τα παιδιά. Προσπαθώ να απαντήσω σε ερωτήσεις με τη σειρά που τέθηκαν. Αν οι Αμερικανοί πολίτες θα τύχουν ίση προστασίες με τους Ευρωπαίους. Αυτή η οδηγία αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες ε, που πέφτουν θύματα εγκληματικής πράξης στην Ευρώπη. Τέθηκε μια ερώτηση και για τις οικογένειες των θυμάτων, για τους οικείους τους. Ε, είπα και προηγουμένως ότι θα επεκτείνουμε την ε, έννοια του θύματος, γιατί πιστεύουμε ότι και οι οικογένειες είναι θύματα μιας εγκληματικής ενέργειας από τη στιγμή που η ενέργεια αυτή αγγίζει ένα μέλος της οικογένειας. Ο κύριος Άλμπρεχτ ε, ρώτησε αν ε, μια οργάνωση μπορεί να εκπροσωπεί το θύμα. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην παρούσα μορφή της πρότασης τουλάχιστον. Εκπροσωπείται το θύμα από μια οργάνωση. Κυρία Γκρισμπέκ, θα σας απαντήσω στα γαλλικά. Καταρχήν, κυρία Γκρισμπέκ, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, EPO, ε, βρισκόμαστε σε φάση ε, συμφωνίας. Έχουμε πολιτική συμφωνία για τις ποινικέ υποθέσεις ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας στις αστικές υποθέσεις γιατί την αλληλένδετες οι ποινικέ με τις αστικές υποθέσεις ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό και αν δεν κάνω λάθος θέσατε και μία ερώτηση για το γεγονός ότι η οδηγία έχει οριζόντιο χαρακτήρα και το πώς θα ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες. Η ερώτηση αυτή συνδυάζεται με προηγούμενη ερώτηση του κυρίου Κίρκοπ. Ο κύριος Κυρκόπ είπε ότι η οδηγία δεν θα υποκαταστήσει το εθνικό δίκαιο. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε ότι εδώ θεσπίζουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα. Και φυσικά υπάρχει ένα επιθυμη... ένας επιθυμητός βαθμός ερμηνείας που επαφίεται στα κράτη-μέλη. Και η προστασία των θυμάτων είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Ο δικός μας στόχος είναι να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα Κάποιες χώρες μπορεί να είναι πιο φιλόδοξες, να προστατεύσουν πολύ περισσότερο τα θύματα. Εξαρτάται από το βαθμό ετοιμότητάς τους, από την οτροπία, από την εθνική ψυχολογία. Δικός μας στόχος πάντως είναι να εξασφαλίσουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα με ένα βαθμό ερμηνείας. Δεν υποκαθιστά λοιπόν η οδηγία το εθνικό δίκαιο. Αναφέρθηκε και το θέμα της θέσης του καθεστώτος του θύματος. Τη νομική θέση του νομικού καθεστώτος. Θα το εξετάσουμε και το θέμα αυτό πιο λεπτομεριακά στη συνέχεια. Νομίζω κύριε Πρόεδρε και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Ελπίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πρόθυμοι για συνέχεια της συζήτησης όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο φυσικά και να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε και πάλι κυρία Λεμπάη. Από ό,τι κατάλαβα, νομίζω ότι έχουμε κλείσει στο θέμα αυτό. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό και ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας. Όχι μόνο για να όχι μόνο την προσπάθεια να περιουσείται στο ουσιώδες, αλλά επίσης το να παράσχεται συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάθε σχόλιο για τον κάθε μέλος της ομάδας που έλαβε το χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση σε ό,τι αφορά διαχείριση του χρόνου. Από ό,τι κατάλαβα προς το παρόν, οι συγητές δεν θέλουν να κάνουν τελική παρουσία, παρατήρηση. Νομίζω ότι καλύπτονται με τις ε, απαντήσεις της κυρίας Λεμπάη. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη κοινή συζήτηση που χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση αφορά σε τρία συνολικά σημεία. Το 7, το 8 και το 9 από κοινού. Καλωσορίζουμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Νότσεν. Παρακαλώ πολύ. Θα λάβετε το λόγο από εκεί, αν θέλετε. We welcome here Madame Knudsen. Καλωσορίζουμε την κυρία Νούτσεν, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Yes, please. Έχετε το λόγο. Βλέπετε ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Η ατζέντα είναι ως συνήθως. έχουν να κάνουν με τα σχετικά θέματα διαδικαστικά, ε, δικαιώματα ποινικά, προσφυγή, δικαστική έρευνα, όλα τα σχετικά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν από τον προτέρων για την κατανόησή σας και για τον πίεση χρόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή να ανατρέξουμε στην μερίσια διάταξη και ξεκινάμε την ε, κοινή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτα στο σημείο 7, που είναι η πράσινη βίβλος. Την πράσινη βίβλο είναι εφαρμογή ενωσιακής ποινική νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης. Σημείο 8. Ανακοίνωση Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο του Συμβούλου για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για μια πολιτική ποινικού δικαίου, κατοχήρωση αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών τη μέσω του ποινικού δικαίου και το σημείο 9 Ανακοίνωση και πάλι τη Επιτροπή για το θέμα εμπιστοσύνη στην πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη, μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρταση. Η κυρία Νούτσε, λοιπόν, από τη Διεύθυνση Ποινική ε, Δικαιοσύνη, διευθύντρια του Τμήματο Ποινική Δικαιοσύνη και χωρί περαιτέρω καθυστέρηση δίνουμε το λόγο στην κυρία Νούτσεν και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση με τα μέλη. Επιμένοντα όμω, εκ των προτέρων, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τον χρόνο εισήγησης κάθε μέλους. Κύριε Νούτσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και συνεκτική όπως και η προϊσταμένη μου, η κυρία Λεμπέη, αλλά επιπροσθέτως νομίζω ότι συμφωνήσαμε να ομαδοποιήσουμε τις τρεις αυτές ανακοινώσεις στην ημερήσια διάταξη αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά, γιατί οι τρεις ανακοινώσεις στην ημερήσια διάταξη δεν αφορούν συνομοθεσία. Αντίθετα με τα σημεία που κάλυψε η κυρία Λεμπάγε, είναι απλώς ανακοινώσεις Και αντιμετωπίζονται από κοινού και συνδέονται με μια κοινή θεματική, που είναι ακριβώς τη αμοιβαία εμπιστοσύνη στα διάφορα πεδία του. Ξεκινώντας λοιπόν με τον πρώτο, που ο τίτλο είναι ακριβώ η ενδυνάμωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνη, και αφορά στην εφαρμογή της ε, ποινική δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τα θέματα κράτησης. Είναι μια πράσινη βίβλος που στόχο έχει να ξεκινήσει μια ευρεία δημόσια διαβούλευση για να εξηγήσει περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ θεμάτων κράτησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Η Πράσινη Βίβλος καλύπτει τα θέματα, ε, επικάλυψη αν θέλετε, μεταξύ αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προδικαστικής κράτησης και η βίβλος θέτει 10 ερωτήματα στο πώ μπορεί να ενδυναμωθεί αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σε αυτή τη φάση λοιπόν δεν υπάρχουν συμπεράσματα, ούτε ε, ζητείται δρα, ανάληψη δράση, θα ήταν πρόωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια αρχική διαβούλευση. Με την βίβλο αυτή πρέπει, θέλουμε να διερευνήσουμε λοιπόν το βαθμό με τον οποίο τα θέματα κράτηση μπορούν να έχουν επιρροή στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατά συνέπεια στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά στην ενδυνάμωση της αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών στα κράτη-μέλη και του να καταστεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πολύ πιο αποτελεσματική όταν ε, έχει αντίκτυπο στην κράτηση. Οι συνθήκες κράτησης ε, ποικίλουν ευρέως τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, οι δικαστές θα ήθελαν να έχουν τη διασφάλιση σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης σε διασυνοριακές υποθέσεις και οι πολίτες επίσης θα ήθελαν να έχουν την εμπιστοσύνη και, την και, το... και να καθυσυχάζονται ότι θα έχουν αντίστοιχες συνθήκες κράτησης όπου και αν βρίσκονται. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί η συνεργασία στα κράτη-μέλη και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά όταν εφαρμόζονται αυτέ τι αρχέ αμοιβαία αναγνώριση. Τα θέματα λοιπόν κράτηση, είτε πρόκειται για προδικαστική κράτηση, είτε για καταδικασμένου, καθώ και τα θέματα διαχείριση φυλακών, είναι θέματα που είναι αμυγό αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχουν όμω πολύ καλή λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσουν τα θέματα αυτά παρά την ισχύ της αρχής της επικουρικότητας. Τα θέματα ε, συνθηκών κράτησης εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας γιατί είναι μια πτυχή των προσωπικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που θα πρέπει να διασφαλιστούν για να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη και να διασφαλίζουν καλή λειτουργία των θεσμών μας και επίσης έχει και προστιθέμενη αξία το θέμα ε, και εμπίπτουν στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που είναι το πρότυπο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα κράτη-μέλη. Όπω επίση γνωρίζετε, το Συμβούλιο, στον οδικό του χάρτη, σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά δικαιώματα, αναφέρεται λεπτομερώ στα ζητήματα κράτηση. Και μάλιστα το Συμβούλιο προσεκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει και να υποβάλει μια πράσινη βίβλο πάνω σε θέματα προδικαστική κράτηση. Και ακριβώ το, ε, η βίβλος αυτή είναι σε ανταπόκριση του αιτήματο αυτού από το Συμβούλιο και η προτινόμενη πρόσβαση σε συνήγορο, όπως παρουσιάστηκε από την κυρία Λεμπάγη, είναι, είναι κομμάτι της του δικού αυτού χάρτη. Επίσης αξίζει να υπενθυμίσουμε εντάχει ότι το πρόγραμμα τη Στοχόλμη επίσης περιέλαμβανε αναφορές στα θέματα αμοιβαίας ε, ε, εμπιστοσύνη και στα θέματα κράτηση. Και επιπροσθέτω, εδώ και αρκετά χρόνια είχε γίνει έκκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματευτεί διάφορα θέματα. Στα πλαίσια ακριβώ και στο ψήφισμα του προγράμματος Στοκχόλμη. είχαν γίνει αναφορές στον κοινό δικαστικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τι συνθήκε κράτηση. Χωρίς την αμοιβαία εμπιστοσύνη στα θέματα κράτησης δεν θα λειτουργήσει σωστά όλος ο μηχανισμός. Γιατί σε ένα κράτος μέλος θα ήταν απρόθυμο να αναγνωρίσει και να επιβάλλει τις ε, απόφαση, δικαστική απόφαση που έχει ληφθεί από ένα άλλο κράτος μέλος και θα παρεμπόδιζε περαιτέρω τη συνεργασία των κρατών μελών, εάν δεν γίνουν προσπάθειε να βελτιωθούν οι συνθήκε κράτηση και να προαχθούν ακριβώ εναλλακτικέ σε ό,τι αφορά την κράτηση. Υπάρχουν τέσσερα εργαλεία αμοιβαία αναγνώριση των όλων δικαστική μα πανοπλία, που μπορεί να διευκολύνουν, αν θέλετε, την ευθυγράμμιση των συνθήκων κράτηση. Το πρώτο είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, που ισχύει και στην προδικαστική διαδικασία και μετά την ε, έκδοση δικαστικής απόφασης. Το δεύτερο είναι η απόφαση πλαίσιο για την μεταφορά ε, κρατουμένων, που είναι ένα καλό παράδειγμα των προβλημάτων που ενδεχομένως ενέχονται στην αμοιβαία αναγνώριση, στο πεδίο της κράτησης. Δεν έχει εισέλθει ακόμα σε πλήρη ε, εφαρμογή Επιπροσθέτως υπάρχουν δύο ακόμα εργαλεία αμοιβαίας αναγνώρισης όπου με τη διάσταση της κράτησης, συγκεκριμένα η απόφαση πάνω σε εναλλακτικά μέτρα κράτησης και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Εποπτείας, Επιτήρησης, που πρέπει να εκδοθούν και να εφαρμοστούν τα κράτη-μέλη το αργότερο μέσα στον επόμενο χρόνο. Κατά τη διάρκεια τη περίοδου αυτή που πρέπει να εφαρμοστούν αυτέ οι αποφάσει από τα κράτη-μέλη, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη τα προβλήματα και του τι συνεπάγονται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κράτηση, του πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματική ε, μεταφορά των ε, νομοθεματημάτων αυτών. Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι η διαδικασία της ε, κράτησης πριν προδικαστικής κράτησης. Το πρόγραμμα Στοχόλμης αναφέρει ότι ποικίλει η περίοδος αυτή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Γενικά, η κράτηση πρώτης ε, ακροματικής διαδικασίας πρέπει να θεωρείται ένα κατεξαίρεση μέτρο στην ομοθεσία των κρατών μέλων και, δεν θα πρέπει, και θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ε, άλλα μέτρα, όπως ε, μέτρα κατοίκων επιτήρησης ή εποπτείας εκτός φυλακής, δεν υπάρχουν. η εποπτειας εκτος φυλακης δεν υπαρχουν η προφυλάκηση ε, σε ορισμένε χώρες δεν περιορίζεται από συγκεκριμένη maximum διάρκεια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η μέγιστη διάρκεια, σε άλλες χώρες η μέγιστη διάρκεια μπορεί να είναι τέσσερα χρόνια. Η άλλη περίπτωση σε σχέση με αυτή την προθεσία είναι όταν υπάρχουν οι, απειρο, απειρο, οι ελάχιστες δυνατές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ε, ε, συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές ε, όταν πρέπει να και το ελάχιστο αν θέλετε θεσπισμένο που υπάρχει για να υπάρξει αυτή η αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη των μελών. Καλύπτονται λοιπόν και τα θέματα διαβούλευσης, γι' αυτό όπως και για άλλα, όπως εναλλακτικέ για την κράτηση παιδιών, καλές συνθήκες κράτησης επίσης, που έχουν σημασία και στα πλαίσια της αποκατάστασης. Τίθενται ζητήματα λοιπόν του πώς κάποιος μπορεί να συντονίσει την εργασία, την, για την παρακολούθηση των συνθήκων κράτησης στα κράτη-μέλη και πώς μπορεί να προαχθεί η δικτύωση μεταξύ των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων που εξετάζουν τις συνθήκες κράτησης, να υπάρξουν καλύτερες συνέργειες, καλύτερες πρακτικές και να επαφήγεται βέβαια η επικάλυψη ε, συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πώς μπορεί να υπάρξει επίσης προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο τι μπορεί να γίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το, το, η όλη προσπάθεια δηλαδή είναι πώς να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των ε, σχετικών δικαιικών συστημάτων. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό απαντήσεων που θα αναλύουν προσεκτικά και θα παρέχουν με ενοποιημένο και συνεκτικό τρόπο κάποια απάντηση για να μπορεί να ε, παγιωθεί κάποια οποιαδήποτε ενδυνάμει μελλοντική δράση στο πεδίο αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά στην ε, νέα ανακοίνωση ποινικού δικαίου που έχει τίτλο προς μια πολιτική ποινικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχήρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Είναι πρώτη φορά που προσπαθούμε να θεσπίσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές στο ποινικό δίκαιο υπό τα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας. Η όλη πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ποινική πολιτικής επί τη βάση των διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνα και βασιζόμενη στην ανάγκη να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ενώ θα γίνονται θα γίνεται σεβαστή μια ε, στιβαρή προσέγγιση σε ό,τι, διαφορά, σε ό,τι αφορά στην προστασία των ε, ατομικών δικαιωμάτων. Είναι μια ανεξελίξη διαδικασία η οποία είναι project. Το ποινικό δίκαιο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο πεδίο σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα με πολύ μεγάλες διαφορές στα σχετικά συστήματα των κρατών μελών. Ως εκ τούτου οι σαφείς και διαφανείς κανόνες είναι εξαιρετικά σημαντικοί σε ό,τι αφορά τη μετώπιση του ποινικού δικαίου. Άρα είναι ένα είδος ε, τεστ, ένας δύο ελέγχου θέσπισης κριτηρίων όταν ε, χρησιμοποιούνται ποινικέ κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια και να παρασχεθεί ένα γενικό πλαίσιο κοδευθυντήριων γραμμών. Είναι πρώτη φορά που γίνεται απόπειρα να γίνει κάτι τέτοιο. Και στόχο είναι επίση να παράσχει μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια σε κοινοτικό επίπεδο, σε αντιδιαστολή με την ε, σχετικό καταγερματισμό που είδαμε σε προηγούμενε περιόδου, πλην την ε, κατακύρωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, βήμα, αλλά ταυτόχρονα χρησιμεύει στην δημιουργία μεγαλύτερης εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών των κρατών μελών. Το νομικό πλαίσιο βέβαια έχει αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας, με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όλα αυτά λοιπόν είναι θετικά κίνητρα στην προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του να δώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά βέβαια η βάση παραμένει ίδια δηλαδή η αρχή της επικουρικότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία εγγυάται η χάρτα και η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ενώ ο συνολικό στόχο λοιπόν είναι η αντιμετώπιση τη κοινή πολιτική, είναι σαφέ ότι η ανακοίνωση εστιάζει στο άρθρο 83.2, δηλαδή στην αποτελεσματική εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών. Ως εκ τούτου το ερώτημα είναι πότε το ποινικό δίκαιο θεμελιώδες για την διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής της ε, κοινοτικής πολιτικής. Πότε υπάρχει έλλειμμα εφαρμογής ε, σε τέτοιο βαθμό που πλέον ε, είναι θεμητές και δικαιολογημένες οι ποινικές κυρώσεις. Ποτέ στο παρελθόν δεν, δεν να εξηγήσουμε με στιματικό τρόπο κάτι τέτοιο. Δεν επισέρχομαι τόσο σε λεπτομέρειε. Η ανακοίνωση δίνει τη μεθοδολογία σε δύο βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να αποφασιστεί κατά πόσο χρειαζόμαστε ποινικέ κυρώσει. Και προκειμένου να αποφασίσουμε επ' αυτού, θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον το μέτρο είναι θεμελιώδε και απαιτεί την επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων στόχων, κατά πόσον η αναλογικότητα ε, ισχύει και εάν περάσουμε όμως το πρώτο βήμα, το κατά πόσον απαιτείται μια ποινική κύρωση, είναι ένα δεύτερο βήμα στη μεθοδό μας. Δηλαδή να αποφασίσουμε τι είδους ε, ποινικά μέτρα μπορούν να υιοθετηθούν. Η συνθήκη προφανώς μας περιορίζει στους ελάχιστους κανόνες ορισμού για τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις και συνθήκες αναγκαιότητας και ε, αναλογικότητας ισχύουν επίσης όταν θέλουμε να αποφασίσουμε τι τύπου κυρώς θα θέλαμε να επιβάλλουμε. Και ο στόχος μας είναι ακριβώς να... Ε, να προσαρμόσουμε και να διαμορφώσουμε τις κυρώσεις σε, συγκεκριμένο σε συγκεκριμένα πεδία και πρέπει να αποφασιστούν και κάποια παιδεία κατά περίπτωση, πολύ συχνά λαμβάνοντα υπόψη εάν υπήρξε προηγούμενη εναρμόνιση σε σχετική κοινοτική πολιτική. Για να πάρουμε συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο βέβαια χρονολογείται πριν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είχαμε περιπτώσει όπου αποφασίστηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε θέματα θαλάσσια και περιβαλλοντική ρήπανση, όπου για πρώτη φορά επιβλήθηκαν κυρώσει. Αυτέ οι οδηγίε ω έχουν τώρα έχουν φτάσει στη φάση που πρέπει να εφαρμοστούν και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγι στην κατάσταση στα κράτη-μέλη. Ήταν τα πρώτα, οι πρώτοι μηχανισμοί οι οποίοι υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία συναπόφηση στο ποινικό δίκαιο. Και νομίζω ότι η συνεργασία που είχαμε την εποχή εκείνη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει κάποιο ένα παράδειγμα στο πώ θα δουλέψουμε και στο μέλλον, όταν θα προκύψουν και άλλε παρεμφενεί περιπτώσει. Το ποινικό δίκαιο, λοιπόν, θα έπρεπε να εστιάσει σε παιδεία όπου υφίσταται ήδη κοινή προσέγγιση. Εν μέρει ακριβώ επειδή το σύστημα κυρώσεων ίσω να μην είναι αποτελεσματικό στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε σε κοινοτικό επίπεδο τον αποτελεσματικό σεβασμό για τους κανόνες που έχουν αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποτεδήποτε υπάρχει έλλειμμα επιβολής ε, του εφαρμογής του νόμου, στην ανακοίνωση αυτή αποφύγουμε θέματα. Για παράδειγμα, θέματα τα οποία συνδέονται με την οικονομική κρίση, προσπαθώντα να ε, επισημάνουμε οικονομικού τομεί όπου ίσω χρειάζεται ε, προστασία ε, των συμφερόντων, για παράδειγμα των φορολογουμένων. Και το κείμενο επισημαίνει και τονίζει τα επικόλθα παιδεία, καταρχά την καταπολέμηση του δόλου, όπου υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του πώς ακριβώς πρέπει να προστατευτούν τα τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον πώς μπορεί να προστατευτεί ο χρηματοοικονομικός τομέας από τις χρηματοκορές και τις κερδοσκοπικές επιθέσεις και τρίτον βασικό ήταν η προστασία του ευρώ απέναντι σε ε, πλαστογράφηση. Ε, ως εκ τούτου σε άλλα πεδία ε, πολιτικής θα θέλαμε επίσης να κάνουμε περαιτέρω ανάλυση για να τοπίσουμε τα συγκεκριμένα πεδία όπου ίσως να απαιτείται ποινικό δίκαιο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει παραβιάσεις σε κατεστημένους κοινοτικούς κανόνες. Και εκεί έχει εντοπιστεί σε μια πρώτη φάση ε, στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές, στους κανόνες περιτελωνίων και το περιβάλλον, την αλία και την εσωτερική αγορά. Αυτά είναι τα πεδία λοιπόν πάνω στα οποία θα συνεργαστούμε και πώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε συγκεκριμένα. Θα δημιουργήσουμε μια ομάδα ειδημόνων που θα εξετάσει μια σειρά θεμάτων συμπεριλαμβανομένης και της ε, συλλογή συγκεκριμένων ε, ε, πιστηρίων. Όπως είδατε και εσείς, πρέπει να έχουμε απόλυτα τα και στιβάρα πιστήρια σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα κράτη-μέλη, το σύστημα κυρώσεων, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ποινικό δίκαιο σε κάθε χώρα μέλος. Θα είναι ζωτική σημασία να έχουμε μια προσέγγιση επί τη βάση πιστηρίων. Θα πρέπει επίσης η ομάδα ειδημόνων στο μέλλον να αντιμετωπίσει μια σειρά θεμάτων όπου υπάρχει ίσως μια ε, ενιαία κατανόηση. Για παράδειγμα, πάτε το θέμα τα ποινική ευθύνη ε, και ε, υπόλογου τα θέματα του νομικά υπεύθυνου, θέματα του πώς ερμηνεύουμε την έννοια της ε, αποτρεπτικής, ε, των αποτρεπτικών, αποτελεσματικών και ουσιαστικών κυρώσεων. Υπάρχει ένα άλλο πεδίο που συνδέεται που αν θέλετε είναι η τομή μεταξύ διοικητικού ε, δικαίου και ποινικών κυρώσεων που θέλουμε να εξερευνήσουμε. Επίσης σκεφτόμαστε να αναπτύξουμε κάποια απλούστερη γλώσσα σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Υπάρχει μια σειρά λοιπόν ε, ε, οδών για περαιτέρω επεξεργασία και διερεύνηση και θέλουμε να εξηγήσουμε το θέμα αυτό ερμηνεύοντας μια σειρά κοινών ενιών σε όλους μας, όπως επίσης και μια σειρά κριτηρίων και κατοφλίων για την εφαρμογή του ποινικού δικαίου. Και σε αυτό έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δομώντας την πολιτική αυτή και θα θέλαμε να συνεργαστούμε στενά μαζί σας στο μέλλον για τις περαιτέρω εξελίξεις. Αυτά περί ποινικού δικαίου. Ήμουν αρκετά σύντομη. Ναι, νομίζω ήμουν το επόμενο θέμα είναι η κατάρτιση. Δικαστική κατάρτιση λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλα αυτά τα τρία ζητήματα υπάρχει συσχέτιση όσον αφορά την, ε, το, το χτίσιμο εμπιστοσύνη. Τώρα, όσον αφορά την κατάρτιση Υπάρχουν περίπου 1,4 εκατομμύρια ε, νομικοί επαγγελματίες στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι οι δικαστές στα κρατημέλη πρέπει να βρίσκονται πάντα ενήμεροι για το κοινοτικό κεκτημένο. Όλοι αυτοί οι φορείς που έχουν σχέση με την κοινοτική νομοθεσία, δηλαδή εισαγγελεί, ε, δικαστέ, δικηγόροι, χρειάζονται να έχουν ελάχιστε γνώσει σχετικά με το κοινοτικό κεκτημένο. Πρέπει να μπορούν να το ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τον κοινοτικό νόμο ε, μαζί με τους εθνικούς νόμους. Έτσι ώστε οι, οι εθνικοί δικαστές να μπορούν να γίνουν πραγματικά κοινοτικοί δικαστές. Αυτό είναι αναγκαίο για να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και πώς σχεδιάζουμε να το καταφέρουμε αυτό. Έχουμε βρει κάποια πρακτικά μέτρα. Όλα αυτά τα μέτρα βασίζονται σε σε κάτι που σε μια συνεδρίαση που κάναμε νωρίτερα φέτος, όπου ζητήσαμε τις απόψεις του κάθε κράτους μέλους. Ένα από τα πράγματα που μάθαμε είναι ότι χρειαζόμαστε ξεκάθαρους στόχους και ξεκάθαρες δράσεις από τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η δικαστική ε, κατάρτιση θα φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε λειτουργική δικαστική λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, είπαμε ότι αρχικά θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε 700.000 ε, νομικούς επαγγελματίες, τους μισούς δηλαδή, να τους δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης μέχρι το 2020. Δεν είναι ευθύνη της Επιτροπής, είναι ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων, των κράτων μελών, των επαγγελματικών οργανώσεων, συμβουλίων, δικηγορικών συλλόγων, δικαστικών σχολών ιδρυμάτων δικαστικής κατάρτισης, των νομικών επαγγελμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Όλοι πρέπει να αναμειχθούν και να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κατάρτιση αυτή. Ζητήσαμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. Ζητήσαμε το εξή πως όλοι οι νομικοί επαγγελματίες θα πρέπει να υποφεληθούν τουλάχιστον μίας εβδομάδα ε, κατάρτισης πάνω στα, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης, προβλέπεται ένα πρόγραμμα ανταλλαγών για δικαστές και εισαγγελίες το 2014. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή είναι το καλύτερο μέσον κατάρτισης όχι μόνο για, πάνω στο κοινοτικό και εκτιμένο, αλλά και στα δικαστικά συστήματα των άλλων κρατών μελών. Φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πόρους που έχουμε και θα θέλαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στους πόρους για την αρχική κατάρτιση, να υποστηρίξουμε προγράμματα υψηλού επίπεδου, προγράμματα κατάρτισης αυτών των επαγγελματιών. Τώρα το κάνουμε προσπαθώντας να βρούμε μέσω των εθνικών προγραμμάτων επίσης μέσα στο μέσα στα εθνικά πλαίσια προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε περίπου 20.000 τέτοιους επαγγελματίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτεραιότητα θα δοθεί σε εισαγγελείς και δικαστές, καθώς εκείνοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την επιβολή της, εθνική, της νομοθεσίας. Και σταδιακά επιθυμούμε όλοι οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου να επωφεληθούν από αυτήν την κατάρτιση. Θα υπάρχει σύνδεση με το πόρταλ δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, τρόποι αξιολόγησης. Θα θέλαμε να κάνουμε επίσης πολύ περισσότερα, έτσι ώστε να προωθήσουμε και τις ε, ιδιωτικές συνεργασίες εκτός από τις κρατικές στον χώρο της κατάρτισης έτσι ώστε να σχηματιστούν μοντέλα λειτουργίας και στον ιδιωτικό και στον ε, δημόσιο τομέα. Έπειτα, στις υπάρχουσες δομές υπάρχουν ήδη αρκετά, αρκετοί ενδιαφερόμενοι, δικαστικές σχολές, ευρωπαϊκοί οργανισμοί, ευρωπαϊκά δίκτυα κατάρτισης, τα οποία θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση που θα συνεχίσει για τα επόμενα 6-7 περίπου χρόνια. Ιδανικά επίσης θα θέλαμε να δούμε κάποιον μηχανισμό αναφοράς. Είναι φιλόδοξη στόχη αυτή, όμως σε κάποιο σημείο θα χρειαστεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αν έχουμε κάνει πρόοδο ως προς τους στόχους μας. Έτσι λοιπόν οι επιτροπές Λίμπε και Τζούρι μας υποστήριξαν πάρα πολύ στο στόχο αυτό. Ελπίζω να συνεχίσουμε να μπορούμε να βασιζόμαστε πάνω, μας, πάνω σας και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νάτσεν. Λοιπόν, επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις τρεις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες και στην παρουσίαση θα αρχίσουμε τώρα μια σύντομη συζήτηση. Έχετε δύο λεπτά ο καθένας. Έπειτα θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Σας ε, ζητώ την κατανόησή σας. Διαφορετικά θα είναι αδύνατο να ασχοληθούμε με όλα τα σημεία της μερίσιας διάταξης, εάν δεν είμαστε σύντομοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κνούτσεν με απόλυτα σαφή και εναργέστο τρόπο μας παρουσίασε συνεκτικά τις τρεις ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τις συνθήκες λοιπόν κράτησης. Διαβάσαμε στην Πράσινο Βίβλο ότι οι διαβουλεύσεις ολοκληρώνονται 30 Νοεμβρίου και θα υπάρξουν στους και άλλες συνεισφορές. Στο πρόγραμμα της Στοχόλμης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη στα οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη σχετική επικάλυψη σε ό,τι αφορά την ύπαρξη πάρα πολλών υπερβολικά μεγάλου αριθμού από τρίτε χώρε θα παρενέβαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και μέσω προγραμμάτων δημιουργίας κάποιας νέας πραγματικότητα ε, ένταξη και ενσωμάτωση προϋπαρχουσών. Αυτό σημαίνει δηλαδή δημιουργώντα και εισάγοντα ε, στα πλαίσια της νέας, των νέων δημοσιονομικών προοπτικών για το 2012-2020. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο είναι το πραγματικό καθεστώς και οι συνθήκες ε, ε, ολοκλήρωσης σε σχέση με τους φιλόδοξους αυτούς στόχους, σε σχέση ακριβώς με την ενσωμάτωση ε, της κρυφής εργασίας παράνομης μετανάστευσης και ιδιαίτερα ακριβώς σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα, πλέον ευάλωτα άτομα, θύματα, δηλαδή τους ανηλίκους. Επίσης, ε, υπενθυμίσατε ότι η προδικαστική κράτηση πρέπει να είναι κατά μέτρο και περιορισμένης διάρκειας. Ποια θα πρέπει να είναι και θα έπρεπε να είναι η θέση της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών του θέματος και ποιες θα πρέπει να ήταν η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιες δραστηριότητες ε, ε ανάκρισης και αναφέρουμε συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα αν θέλετε, τις δεχόμενες ε, υποκλοπές, ε, τηλεφωνικές υποκλοπές γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ε, ε, απέτηση να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και προδιαγραφές και σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση ιδιαίτερα του οργανωμένου κλίματος. Ευχαριστούμε. Κύριε Σκάντς. Ε, κυρία Κίνγκα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, μια και υπάρχει δυνατότητα να μιλήσω στα ογγρικά, να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και επίβολο πρόγραμμα και για να το θέσουμε σε εφαρμογή χρειαζόμαστε και την ανακοίνωση και την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια αυτή τη στιγμή περισσότερα ερωτήματα έχουμε παρά απαντήσεις. Αναφέρθηκε πολλάκις το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται αρκετά το πλαίσιο που υπάρχει στα κράτη-μέλη. Και νομίζω τα δύο έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζουν κάποια μέσα και εργαλεία που θα ενισχύσουν τη συνεργασία και θα εκμεταλλευτούν τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς, ώστε με κάποια ελάχιστα πρότυπα να αισθανθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι είναι πραγματικά Ευρωπαίοι πολίτες και τη χάνουν προστασίας παντού. Θα ήθελα να θα σε κάτι που κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την εφαρμογή αυτών των ελάχιστων κανόνων. Έχουμε καταρχήν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλες τις χώρες μέλη. Υπάρχει και το θέμα της ηλικία, από ποια ηλικία και μετά μπορεί κανείς ε, να διωχθεί ποινικά γιατί έχουμε κάποια δικαιώματα που θα πρέπει να έχουν προστασίας και στο τομέα της κράτης υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις συνθήκες. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, έχουμε διάφορα στατιστικά στοιχεία που μας δείχνουν ότι οι μισοί δικαστές εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρίζονται ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση για το κοινοτικό δίκαιο. Νομίζω ότι ε, καλό θα ήταν να αυξηθεί ο αριθμός ε, των ε, υπαλλήλων του νόμου που παρακολουθούν τέτοια επιμόρφωση. Κύριε Λάτφορτ, νομίζω ότι είναι πήγον να ασχοληθούμε με το θέμα της κράτησης και χαίρομαι για τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ενώ δεν έχουν καταδικαστεί επίσημα, κρατούνται χωρίς λόγο μήνες για να μην πω και χρόνια. Αναφέρθηκατε στην περίπτωση μιας χώρας που είχε για τέσσερα χρόνια προδικαστική κράτηση έναν ύποπτο. Χωρίς ε, καμία καταδίκη, χωρίς καμία δικαστική απόφαση, χωρίς καμία απόδειξη ενοχής και μάλιστα η κράτηση αυτή πολλές φορές γίνεται σε απάνθρωπες συνθήκε. Το ανθρώπινο κόστος μιας τέτοιας παράνομης κράτησης ε, μπορεί να είναι τεράστιο. Έχουμε και περιπτώσεις που αλλοδαποί υπήκοοι ε, υφίστανται πολύ περισσότερα δεινά από τους, ε, από τους ημεδαπούς ε, γιατί πολλές φορές κρατούνται προδικαστικά άδικα ενώ θα μπορούσαν να τύχουν άλλων μέτρων πριν τη δίκη τους και κρατούνται ακριβώς επειδή δεν έχουν επίσημη διεύθυνση παραμονής στην χώρα στην οποία διαμένουν και της οποίας δεν είναι υπήκοοι. Επίσης, ε, πολλές φορές γίνεται κατάχρηση και του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως. Γιατί δεν τηρούνται αυστηρέ προποθέσει του Ευρωπαϊκού Εντάλματο ε, Συλλήψεω και μερικοί παραδίδονται ε, σε τέτοια διαδικασία ενώ δεν υπάρχει επικείμενη δίκη. Όταν δεν είναι καν όριμη κατάσταση για μια δίκη σε συγκεκριμένη χώρα. Αυτό είναι το της έρευνας κανονικά. Και κανείς μπορεί προδικαστικά να βρεθεί στο κρατητήριο ένα χρόνο μπορεί να βρίσκεται στο κρατητήριο και μετά ένα χρόνο περιμένοντας την ε, εγγύηση ή την ε, απελευθέρωση. Επίσης, ε, ελπίζω και το ένταλμα επιτήρησης να τηρηθεί όταν τεθεί σε ισχύ, γιατί τα χρήσιμο μέτρο. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι χρήσιμη, γιατί αποκλείεται αμοιβαία αναγνώριση όταν έχουμε τόσο κατάφορες ε, παραβιάσεις ε, ε, σε συνθήκες κράτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τόσο μεγάλες διαφορές. Ο κύριος Δεγιόγχα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδυάζεται και με το αντίστοιχο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα επίκειται και σχετική δημόσια ακρόαση στην οποία συμμετέχω ενεργά. Ποινικό δίκαιο. Το θέμα είναι θα έχουμε μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση, θα έχουμε ένα είδους πανευρωπαϊκό πλαίσιο για το ποινικό δίκαιο ή μήπως ε, λόγω των διαφορών ε, θα επιλέγει κανείς το υπιότερο ποινικό δίκαιο. Να μην καταλήξουμε σε ποινικό τουρισμό, σε φρονιστικό τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν επικρατήσουν σημαντικές διαφορές, αυτό θα συμβεί τελικά. Ελπίζω να αποφευθεί αυτό το σύστημα να χρησιμοποιούν και να, εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες ε, τις διαφορές μεταξύ των ποινικών δικαίων των χωρών μελών. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κοινά κριτήρια, για παράδειγμα υπογραφή ε, διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. Νομίζω ότι αυτός είναι αρκετός λόγος ε, να προωθήσει τέτοιου είδους ε, ευρωπαϊκή προστασία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχουν κοινοί γνώμονες και κριτήρια. Σημαντικό πράγμα είναι η συνέπεια. Αλλά πώς θα γίνει ο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην κάτω χώρες έχουμε Υπουργείο Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο, αλλά τι γίνεται σε περίπτωση που η παραβίαση είναι παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας ποια διεύθυνση θα είναι αρμόδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε συντάξει σχετικό ψήφισμα, αλλά φαίνεται ότι και η αρμόδια Επιτροπή Μάλμστρομ δεν δίνει προτεραιότητα σε τέτοια θέματα. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομη. Είπατε πω οι εγκληματίε δεν θα πρέπει να επιζητήσουν τι καλύτερε συνθήκε κράτηση, όμω πρέπει να υπενθυμίσω ότι δεν είναι όλοι οι κρατούμενοι εγκληματίε, κάποιοι είναι και αθώοι. Και όταν κάποιο συλλαμβάνεται και πραγματικά είναι ένοχος, τότε καταδικάζεται, δεν, δεν τον εκδικούνται. Στόχος επίσης πρέπει να είναι τα, οι ποινέ αυτές να είναι έτσι, να είναι τέτοιες ώστε να μην επαναληφθεί το αδίκημα αυτό πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ενσωματώσουμε στην όλη διαδικασία. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικέ λύσεις για λιγότερο σημαντικά δικήματα από την φυλάκηση. Όσον αφορά την εναρμόνιση και την, την ενσωμάτωση της, κοινωνική, της κοινοτικής νομοθεσίας, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και όσον αφορά τη δικαστική κατάρτιση τώρα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι όμως κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσει έναν δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε όλους τους τομείς. Ελπίζω όμως αυτή η ανακοίνωση να οδηγήσει σε επικοδομητικές συζητήσεις στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νούτσε, να έχετε το λόγο. Ή, ε, όχι, υπάρχει και ο κύριος Μπρόγκς που θα ήθελε να μιλήσει. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Μάλιστα. Πιστεύω πως ένας από τους λόγους που, καθυστερούν, που, που υπάρχουν καθυστερήσεις στις προδικαστικές διαδικασίες είναι ότι οι προανακρίσεις κρατάνε τόσο πολύ. Οι προανακρίσεις σε περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με τρομοκρατία περιορίζονται στις τέσσερις ημέρες. Ίσως το Ίσως το υπηρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο να έχει κάτι να διδάξει στο βρετανικό ποινικό δίκαιο. Κύριε Ακνούτσεν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας. Έχουμε κάποιο χρόνο να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι, σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες στο μέλλον να το συζητήσουμε αυτό. Αυτό που λαμβάνω από τα σχόλιά σας είναι ότι το ζήτημα της αμοιβαίας αναγνώρισης είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουμε νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα καθόλου και εν μέρει αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολείται η Πράσινη Βίβλος. Μπορούμε να το εξετάσουμε αφού δούμε τις απαντήσεις σας. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα στα πλαίσια της αμοιβαία αναγνώρισης να, κάνουμε, να αναλάβουμε περαιτέρω δράσεις. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, υπάρχουν ήδη κάποια προγράμματα, υπάρχουν κάποια χρήματα μπορούν να διατεθούν για την κατάρτιση, για την εκπαίδευση. Επίσης, περιμένουμε να δούμε και τι θα προκύψει από το πολυεθνικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο. Ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα φυσικά βρίσκεται στο κέντρο της ε, δουλειάς μας, γιατί πρόεδρος ε, Ρέντινγκ αντιπροσωπεύει και αυτό και την ποινική δικαιοσύνη. Και είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά που κάνουμε. Μπορούμε μόνο να θέσουμε ελάχιστους κανόνες. Έτσι είναι τα πράγματα. Και ακόμα και σε αυτό το τομέα όμως δεν έχουμε ιδιαίτερες αρμοδιότητες στον τομέα της κράτησης. Όσον αφορά για εναλλακτικέ λύσεις ε, για την κράτηση, πιστεύω ότι υπάρχει μια απόφαση πλαίσιο για ε, εντολή παρακολούθησης που θα παρέχει περισσότερες δυνατότητες στα κράτη-μέλη ε, από την ηλεκτρονική παρακολούθηση των φυλακισμένων. Όσον αφορά την δικαστική κατάρτιση, που αρκετή κάνατε λόγο για αυτό το θέμα, εδώ έχουμε ήδη αναφέρει και καλύψει κάποια πράγματα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, αυτά για τα τρία σημεία προς το παρόν. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Πλησιάζουμε το τέλος αυτής της μακράς συνεδρίασης. Κυρία Κνούτσεν, ανυπομονούμε να ακούσουμε περισσότερα. Τώρα, το τελευταίο σημείο που αφορά την έκθεση που συνέταξε η συνάδελφός μας, κυρία Σιλβί Γιόμ, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας στα κράτη-μέλη, την αναδιατύπωση. Αυτό το σημείο έχει ήδη συζητηθεί. Έχει ήδη γίνει συζήτηση, όχι πολύ καιρό πριν, πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία συζήτηση και η συγγήτρια κυρία Γκυγιόν, η Επιτροπή και οι σκιώδες συγγητής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το έγγραφο αυτό. Αυτό που προτείνω τώρα είναι το εξή. Εάν η Μαντάμ Κιγιόν ήθελε να μας συνοψίσει την ισχύουσα κατάσταση ή αν κάποιος θα ήθελε να συνεισφέρει κάτι παραπάνω, να κάνει ένα παραπάνω σχόλιο ή μια ερώτηση προς την Επιτροπή, θα χρησιμοποιήσω το χρόνο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλήσαμε ήδη την περσμένη εβδομάδα για το θέμα αυτό. Έχουμε κάνει λίγο τα πράγματα βιαστικά, είναι λίγο κρίμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. Όντω είχα την ευκαιρία να θέσω κάποια ερωτήματα, στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω θα έχει την ευγενή καλοσύνη να απαντήσει, κατά τρόπο που και άλλοι είχαν θέσει κάποια ερωτήματα. Θα ήθελα λίγο να μα δώσει την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στην έκθεση αυτή, πάνω στο θέμα αυτό. Καλώς. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόσδεκτη να μας ε, ενημερώσει για την κατάσταση όσο έχει. Αλλά ίσως, όπως πρότεινε η κυρία Γκυγιόμ, μπορώ να ακούσουμε την κυρία Γκάν από την Επιτροπή, τον κύριο Σόστακ από το Συμβούλιο και μετά βλέπω κάποια χέρια κάποιων που θα θέσουν ερωτήματα. Να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαστόμα της κυρίας Γκάν. Ή το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να κάνει κάποια σύνοψη. Να, ωραία, το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και είναι χρήσιμο αν θέλετε και στην για την Προεδρία να δώσουμε μια ενημέρωση ότι συμβαίνει, πώς έχουν τα πράγματα. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση του κειμένου το Σεπτέμβριο από το Συμβούλιο η Προεδρία δούλεψε σε κάποιες συμβατικές προτάσεις, τις οποίες πρότεινε στην ομάδα εργασίας τον Οκτώβριο. Εργαζόμαστε τώρα πάνω σε μια σειρά συμβαστικών ε, προτάσεων σε άλλα άρθρα, εν ώψη της ε, Συνόδου της ε, Ομάδος Εργασίας για το Άσυλο τον Νοέμβριο. Είναι δύσκολο το κείμενο αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά πολύπλοκο τεχνικά. Χρειάζεται πάρα πολλούς χρόνους, λοιπόν για να περάσουμε λεπτομερώς όλες τις διατάξεις. Η πρώτη ανάγνωση του κειμένου στην ομάδα εργασίας απέτησε τέσσερις ολόκληρες εργάσιμες ημέρες. Και είναι επίσης πολύπλοκο για τις ορισμένες ε, περιπτώσεις έρχεται και διηγεί τα γενικό διαδικαστικό δίκαιο στα κράτη-μέλη και επομένως ο συμβασμός πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο να ξεδεθεί. Όμως η δύσκολη αυτή συζήτηση έχει υποβοηθεί καταρχάς από τις αλλαγές που έχει εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμβαστικές προτάσεις και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις αλλαγές που έχουν εισαχθεί σε ό,τι αφορά τα θέματα ε, νομικής αρρωγής. Και δεύτερο, στα θέματα τα οποία έχουν εισαχθεί είμαστε λιγότερο ουσιαστικοί, αλλά θεωρούμε παρόλα αυτά ότι οι αλλαγές που έχουν εισαχθεί είναι μάλλον επικοδομητικές στην εργασία της ομάδας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή συγγνώμη, πήξε εξαιρετικά επικοδομητική. Η δεύτερη φάση λοιπόν είναι ένα δεύτερο πακέτο συμβαστικών προτάσεων που θα παρουσιάσει στην ομάδα εργασίας η Επιτροπή. Καλώς. Ας ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους ε, Μποσούτιλα και Άλβαρο που θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Ναι, μιλώ εκ μέρους του ΕΛΚ του σκιώδου συγητή του ΕΛΚ επί του θέματο αυτού. Προφανώς ε, συμμερίζομαι τον χαιρετισμό του συναδέλφων για την αναθεωρημένη αυτή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δούμε σωστή κατεύθυνση και επίσης επιχαίρω για τη νέα αυτή ορμή που έφερε η Πολωνική Προεδρία στο θέμα του ασύλου. Εντάχει λοιπόν κάποιες θετικές πτυχές που θέλει να επισημάνει το ΕΛΚ από την τρέχουσα κατάσταση της βελτιώσης σε ό,τι αφορά την παροχή νομικών συμβουλών και προφόρησης, τις επιταχυμένες διαδικασίες και επίσης την, ε, τις νέες διαδικασίες, αλλά επίσης θέλω να επισημάνει κάποιες αρνητικές πτυχές που εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μας ε, βάζουν σε μάλλον δύσκολη κατάσταση. Ε, να, και πολύ μεγάλης απόστασης από τον κανονισμό. Καταρχάς ε, της ε, αυτόματης διαδικασίας ανάκλησης. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κατάχρηση και επομένως τα δικαστήρια στα κράτη-μέλη θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκφραστούν πάνω στην ε, επιρροή της ε, άρσης και της δυνατότητας ε, ανάκλησης της. Επίσης, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια αιτήματα με επιταχυνόμενο τρόπο, εκτός αν πρόκειται για την τρίτη ή η τρίτη ή η ύστερη ευλογή είναι υπερβολική. Θεωρούμε ότι η επιταχυμένη διαδικασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη από τη δεύτερη αίτηση κιόλα ε, για τη χορήγηση ασύλου. Το τρίτο και είναι σημαντικό, το γνωρίζει αρκετά καλά η Σιλβή Κιγιόμ. Αναφέρω ένα τελευταίο σημείο εδώ πέρα εν ώψη των, ε, των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων. Είναι το θέμα ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Δεν πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να βάζουμε σε κουτάκια τους ανθρώπους ως ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες κάτω από μια συγκεκριμένη ονοματολογία ή κριτήρια όπως είναι η ηλικία ή σεξουαλικός προσανατολισμός. Ο παράγον της ηλικία δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αυτόματα ένα άτομο με ειδικέ ανάγκες. Μπορούμε να έχουμε ένα κάποιον προχωρημένης ηλικία χωρίς να έχει κάποιες ιδιαίτερες ειδικέ ανάγκες και κάποιον σχετικά νεότερο που ίσως να έχει ειδικέ ανάγκες. Δεν θα έπρεπε λοιπόν απλώς να ε, ταξινομούμε τα άτομα ως άτομα με ειδικέ ανάγκες, αλλά μάλλον να κοιτάμε το άτομο ως προσωπικότητα και ατομικά, μεμονωμένα. Σταματώ με αυτό προς το παρόν, λόγω των χρονικών περιορισμών, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που θα, το ΕΡΚ θέλει να επισημάνει ακόμα. Ευχαριστώ κύριο Σάλβαρο. Ευχαριστώ. Όπως και ο Σάιμον, Έχω και εγώ την τιμή να την προσωπεύω τη συνάδελφό μου κυρία Χίρς εδώ. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Χίρς τις έστειλε και γραπτά. Πρέπει να υπάρχουν στη Γραμματεία και στην Κομισιόν οι ερωτήσεις αυτές. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω στο όνομά της, καταρχάς στην Κομισιόν, στο άρθρο 23. Το Κοινοβούλιο έκανε λόγο για καταρτισμένους ειδικού ως, ε, με την λειτουργία του συνοδού. Γιατί στα άρθρα 19 και 25 δεν αναφέρεται αυτό. Έπειτα, στο άρθρο 21 αναφέρονται οι νομικές και τεχνικές απόψεις. Η συνάδελφός μου εδώ θέλει να ρωτήσει γιατί δεν αναφέρονται και οι ανεξάρτητες ανεξάρτητες κρατικές θέσεις. Όπως προείπα, οι ερωτήσεις υπάρχουν και γραπτά. Εγώ κάνω απλά μία σύνοψη. Ψήφισμα του Κοινοβουλίου του, το 2009 έκανε κάτι πάνω σε αυτό, τώρα βρισκόμαστε σε μία στάσιμη περίοδο όσον αφορά την αναγνώριση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μίλησε για μια ύστερη φάση όπου θα μπορούσε να εξεταστεί το θέμα. Ε, Η κυρία Oui, την ευκαιρία να πω στο Σιλβί Γιώμ κάποιες συγκεκριμένε παρατηρήσεις ε, εκ μέρου της ομάδας μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάνω στο θέμα του ορισμού της αρμόδιας αρχής και της υπεύθυνη αρχής για να αποφευχθεί πάση θυσία να δοθεί κάποια, να αποφανθεί και να δώσει κάποια απόφαση, κάποια αρχή άλλη απέναντι της αρμόδιας. Ε, η πρόταση δεν αποσαφηνεί στο σημείο αυτό. Μάλλον κινείται αντίθετα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αναφέρουν συγκεκριμένα στο άρθρο 4.2 πολύ μεγάλη προσοχή επαγρύπνησης θα πρέπει να δοθεί και στη διαδικασία ε, σε ό,τι αφορά να ακολουθούμε τη διαδικασία στα σύνορα. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τα καράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν πέραν των 72 ωρών την επεξεργασία του αιτήματο ε, πολιτικού ασύλου. Είναι μια γενική προβληματική στα σύνορα, όπου ακριβώς εκεί ε, απαιτούνται και είναι δυνατές οι επιταχυμένες διαδικασίες. Επιχαίρω ε, βεβαίω και χαίρομαι για το ότι προτείνονται συγκεκριμένε διαδικασίε ε, για τους ανηλίκους. Είναι προφανώ εξαιρετικά θετικό αυτό. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέρχεται με την έννοια της σίγουρη χώρα. Βρήκαμε κάτι σχετικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε ικανοποιηθεί από όλε τι πολιτικέ ομάδε και είναι πραγματικά εκπληκτικό το ότι μας δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε τόσο λίγες κοινέ απόψεις. Η επιταχυνόμενη διαδικασία ναι, είναι δύο νέες περιπτώσεις. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι στο κοινοβούλιο αυτό το βρήκαμε ε, να παράταθεί και να επιμηκυνθεί ο κατάλογος αυτός. Κατά μένα αυτό είναι προβληματικό. τέλος πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το νομικό ζήτημα, την παρουσία των μη κυβερνητικών οργανισμών στο κέντρο κράτησης που δεν αναφέρονται πλέον άμεσα και τέλος το ζήτημα της γλώσσας γιατί ο φορέας θεμελιωδών δικαιωμάτων μας ζητά να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που θα γίνουν θέμα των θεμάτων αυτών. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα μπορούσαμε να ακούσουμε την κυρία Γκάν, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, που θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω να απαντήσω στην πληθώρα ερωτήσεων που τέθηκαν. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την παράταση της προθεσμίας για την εγγραφή των αιτήσεων. Από 72 ώρες περάσαμε σε 7 ημέρες σε περίπτωση μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Επίσης, ε, αναλάβαμε τη δέσμευση να δώσουμε πρακτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα του κάθε κράτους μέλους. Έχω την αίσθηση ότι το πιο σημαντικό είναι τα ίδια τα κράτη-μέλη να ικανοποιήσουν τις άμεσες ανάγκες των αιτών των άσυλων σε ό,τι αφορά την υποδοχή τους και αυτό είναι προτιμότερο από το να οριστικοποιήσουν τις διοικητικές διατυπώσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτοί, αυτές οι 7 ημέρες υπάρχουν, αυτή η διορία. Και φυσικά αυτή η παράταση της διορίας θα πρέπει να είναι προσωρινή και δικαιολογημένη και υπάρχει πρόσβαση στις διαδικασίες και τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο που θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που είχε θέσει την προηγούμενη φορά η κυρία Κιγιόμ για την δυνατότητα αναβολής της λήψης απόφασης σε περίπτωση αβεβαιότητας της κατάστασης στη χώρα προέλευσης του ετούντος και τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα νομικό κενό ε, η Τζιν Λάμπερτ αποουσιάζει, αλλά είναι σημαντικό να γίνει εδώ συσχετισμός με την οδηγία ε, για τους χαρακτηρισμούς. Όπως ξέρετε, η τωρινή οδηγία του 2004 προβλέπει δυνατότητα απόρριψης της αίτησης, ακόμη και αν υπάρχουν μόνιμα εμπόδια με την επιστροφή. Και χάρη στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλείψαμε αυτή τη ε, διάταξη, κάτι που συνιστά πρόοδο κατά τη γνώμη μας. Ακόμη και όταν είναι προσωρινά όμως τα εμπόδια, καλό είναι να υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μπορούν να αναβάλουν λίγο την λήψη απόφασης. Πάντως το πρωταρχικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου ό,τι αφορά τις διορίες ε, στις άσυλο είναι το 6 συν 6 και όχι το 6 συν 1. Δηλαδή, 6 μήνες συν 6 μήνες. Ξέρετε ποιες ε, είναι, ποια είναι η κρατούσα γνώμη στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά και εκεί θα υπάρξει διελκυστίδες διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του ΕΛΚ, ευχαριστώ καταρχήν την αναγνώριση των θετικών στοιχείων που επιφύλαξε η ομάδα του ΕΛΚ στην πρόταση. Με ενδιαφέρουν φυσικά και οι παρατηρήσεις για το ανασταλτικό, αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα που μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση αυτής της διάταξης. Και αυτό θα είναι σημαντικό στοιχείο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο σκελών της νομοθετικής αρχής. Πάντως και το Κοινοβούλιο φυσικά θα ενδιαφερθεί για την ε, τήρηση των αρχών του κοινοτικού δικαίου, του νοσιακού δικαίου, καθώς και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό το πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τα, τις επανειλημμένες αιτήσει, αυτό το θέμα είναι δύσκολο και από τεχνική άποψη, αλλά θα διαβιβάσουμε στην Επιτροπή σας ένα μικρό διάγραμμα και στο Συμβούλιο για να γίνει κατανοητή η δομή της τροποποιημένης πρότασης ό,τι αφορά τις επανειλημμένες αιτήσει. Νομίζω ότι με την πρότασή μας διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη, τηρώντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα εξέτασης των επιτόπιων αιτήσεων ασύλου και χρειάζεται και ένας μηχανισμός για την περίπτωση αυτή. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με ειδικέ ιδιαίτερες ανάγκες, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι αυτές οι ιδιαίτερες ειδικέ ανάγκες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μετά από εξατομικευμένη εξέταση των συνθήκων. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις κυρίας Χίρς, το θέμα του ορισμού των αρμόδιων εθνικών αρχών ε, που γίνονται δεκτές στο νομικό συμβούλιο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των εθνικών συστημάτων για τα θέματα αυτά. Εμείς ε, προτιμούμε μια διατύπωση ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο δυνατόν δυνατό περισσότερες καταστάσεις με τον ορισμό αυτό. Μια και βλέπω τον πρόεδρο σας ε, να αδειμονεί. Ολοκληρώνω και περιμένω και ε, διμερώς τις προτάσεις για επαφές. Δεν είναι ο πρόεδρος που αδειμονεί, οι διερμηνείς είναι που αδειμονούν και παρόλα αυτά μας ε, παραχώρησαν παράταση του ωραρίου τους κατά ένα πεντάλεπτο. Ακούσαμε λοιπόν και την Πολωνική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωβουλευτές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Κυρία Κιγιόμ, αν θέλετε ένα καταληκτικό σχόλιο ή όχι. Δεν χρειάζεται. Πολύ ωραία. Οπότε τελειώσαμε. Τελειώσαμε προς το παρόν αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Λίγη τη συνεδρίαση.